Συνάδελφοι, περιμένουμε ένα-δυο λεπτά για τους κοιόδης ηγητές για την έκθεση του κυρίου Ζόγκορ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την ε, γνωμοδότησή του. Θα περιμένουμε δύο-τρία λεπτά, λίγη υπομονή και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Απλώς ε, ενημερωτικά για την μικρή καθυστέρηση. Good afternoon, colleagues. Um, uh, Καλησπέρα σα, ε, συνάδελφοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τη συνεδρία. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 1, την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, συγκρίνεται Τώρα, γλωσσικό καθεστώ, δεν θα υπάρχει διερμηνία σήμερα στα κροατικά και στα ιρλανδικά. Η υπενθύμηση σήμερα θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 5 παρα 20. Παρακαλώ λοιπόν να έχετε τις κάρτες μαζί σας για την ψηφοφορία στις 5 παρα 20, 16 και 40. Ξεκινάμε τώρα με το πρώτο σημείο, σημείο παριθμών 3, σχέδιο γνωμοδότης του κυρίου Σόγκορ για την ε, έκθεση για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια ένωση της δημοκρατικής αλλαγής. Οι εισαγωγικά συνέδελφοι, να σας πω ότι στις 24 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια του 2017. Η έκθεση αυτή ε, δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια και καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες ε, που λαμβάνονται για να προωθήσουν και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η Επιτροπή Αναφερών ε, είναι επί αρμόδια για την έκθεση, για την ηθαγένεια και η ΛΥΜΠΕ είναι συνδεδεμένη επιτροπή βάσει του άρθρου 54. Έχουμε λοιπόν οριζόντιες επιμερισμένες αρμοδιότητες και αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απειλές ασφαλείας στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάση αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών στο εξωτερικό και προστασία και υποστήριξη των θυμάτων, εγκλημάτων και ε, μαρτύρων. Ο κύριο Σόγκορ θα μα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότηση. Παρακαλώ λοιπόν κύριε Σόγκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε βάσει της συμφωνίας μεταξύ των Προέδρων ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ΠΕΤΗ που περιλαμβάνεται στην έκθεση ε, θα υπάρχει επιμερισμένη αρμοδιότητα ε, με εξαίρεση τα θέματα του σημείου 5 της έκθεσης που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας στον τομέα τη δικαιοσύνη και των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει αμοιβές εμπιστοσύνη, προστασία των Ευρωπαίων πολιτών στο εξωτερικό και προστασία και υποστήριξη των θυμάτων θυμάτων εγκλήματος και των μαρτύρων. Επειδή υπάρχει όρια ε, στους χαρακτήρες, επειδή είναι γνωμοδότηση, ασχολούμαστε αποκλειστικά σχεδόν με αυτά τα θέματα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΛΥΜΠΕΣ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τα εξής. Πρώτον, η ανάγκη να εφαρμόσουμε ταχύτατα το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, ώστε να νιώθουν ασφαλείς οι πολίτες και ότι προστατεύονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, τη σημασία της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της αντιμετώπισης της, ε, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω της ζωφερής πραγματικότητας ε, που ε, βιώνουμε, το γεγονός δηλαδή ότι οι δράστες των πιο πρόσφατων επιθέσεων ήταν Ευρωπαίοι πολίτες και επίσης να υπάρχει μόνιμη προστασία για τους Ευρωπαίους πολίτες στο εξωτερικό και να είναι πιο αποτελεσματική και να υπάρχουν και κατεπήγοντα ταξιδιωτικά έγγραφα. αυτά τα λίγα στοιχεία βέβαια δεν επιτρέπουν παρά να δούμε τα βασικά στοιχεία και γι' αυτό ακριβώς το λόγο με τη βοήθεια των σχεδόν εισηγητών θα ήθελα να επεκτείνουμε την γνωμοδότηση και σε άλλους τομείς. σε Αυτή τη στιγμή ε, συντάσει το γραφείο μου κάποιες τροπολογίες, τις οποίες θα δώσω στους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές για να μπορέσουν να τα λάβουν και αυτοί υπόψη τους στις εργασίες τους και ελπίζω να μπορέσουν να τις προσυπογράψουν κιόλα. Οι τροπολογίες αυτές θα αναφέρονται στα εξή θέματα. Όσον αφορά το θέμα της πρόθεσης της ισότητας όλων των Ευρωπαίων πολιτών, την ανάγκη να υπάρχει αναφορά στις μειονότητες ε, στο άρθρο 2 της συνθήκης ε, και ε, σε ένα καθεστώς μετά την ένταξη θα πρέπει να εγγυόμαστε την ισότητα των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές τις μειονότητες, να ενισχύσουμε την πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα και ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει σεβασμό τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίση, πρέπει να σταματήσουν οι διακρίσει για του ΛΟΑΔ και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά του και επίση να άρουμε όλα τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία για να μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά του χωρίς προβλήματα. Και επίσης την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις αισθηματικές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν κάποιοι πολίτες στις χώρες τους, καθώς επίσης και την απέλασή τους και την εκδίωξή τους όταν ε, ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης ε, μετακίνησης και διαμονής σε άλλο κράτος μέλους. Τώρα, όσον αφορά τους απάτριτες. Ε, το γεγονός ότι αποκλείονται από την προστασία που προσφέρει η ηθαγένεια και τα ωφέλη της ευρωπαϊκής ηθαγένειας δεν επιτρέπουν σε κάποιους ανθρώπους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και βρίσκονται σε ε, δεινή κατάσταση, κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το Brexit, θα ήθελα να αναφέρω την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμα για το Brexit, τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να εγκατασταθούν και να ζουν ε, και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη των 27 θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι κάποια θέματα και θέματα τα οποία ελπίζω να αναπτύξουν και οι ισχυώδει εισηγητές και προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστα από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ε, έχει το λόγο για να εκφράσει την ε, άποψη του συναδέλφου του. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Βάιντενχολτς, ο συνάδελφός μου που είναι αρμόδιος, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα εδώ και γι' αυτό με παρακάλεσε να παρουσιάσω την ε, δική του την γνωμοδότηση. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω είμαι ευγνώμων ε, που συντάσσεται αυτή η έκθεση. Η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κομβική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για να μπορούν οι πολίτες να ταυτιστούν με την Ευρώπη. Ο πολίτης λοιπόν έχει τη ε, δυνατότητα να θεωρεί τον εαυτό του κυρίαρχο. Η νομοποίηση προκύπτει από τις συνθήκες. Ε, για τη γνωμοδότηση λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το ερώτημα το πώς ακριβώς μπορούμε την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την ενισχύσουμε περαιτέρω. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην προστασία του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κατά τη γνωμοδότηση, ε, κατά την άποψή μου πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο στην γνωμοδότηση είναι να υπάρξει ε, εξέταση του ψηφιακού περιχωμένου περιεχομένου της ψηφιακής δυνατότητας να ενισχυθεί αυτή η ελευθερία της ε, ψηφιακής ε, χρήσης και για να μπορούν οι πολίτες ε, να χρησιμοποιούν και να καταφεύγουν στα δικαιώματά τους πρέπει καταρχήν να τα γνωρίζουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακόμα δυστυχώς δεν υπάρχει αποτελεσματική προξενική προστασία. Οφείλουμε λοιπόν να μεριμνήσουμε, να είναι σωστά ενημερωμένοι οι πολίτες για να μπορούν και να απολάβουν τα δικαιώματά τους. Παράλληλα όμως δεν διακυβεύεται μόνο το θέμα της ε, ενημέρωσης, αλλά πρόκειται και για την επέκταση της Ιθαγένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συναφών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διαλόγου με τους πολίτες δεν φτάνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αμυγή σε δημοκρατική μεταρρύθμιση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή είναι ο μόνος άμεσα εκλεγόμενος θεσμός, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν οφείλει να ε, διαδραματίσει πιο θαραλέο και ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά την περαιτέρω επέκταση αυτών των δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε τον κύριο Κιώστα και αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο από τους συναδέλφους, α, όχι, θέλει το λόγο ο κύριος Μπάτμου. Δυστυχώς όμως ε, δεν ακούει. Α, το μικρόφωνο. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατική συμμετοχή. Ένας τρόπος ε, που μπορεί κανείς να το κάνει και ίσως αυτό μπορείτε να το λάβετε υπόψη στην έκθεση είναι ε, οι ευρωβουλευτές που εκλέγονται και αυτοί άμεσα να μπορούν να ψηφίζουν για μεμονωμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι να υπάρχει μία ε, ψηφοφορία συλλήβδη, unblock. Εξάλλου, αν πραγματικά θέλουμε να ακολουθήσουμε το δημοκρατικό δρόμο για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, θα πρέπει να πούμε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι τα άτομα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν υπουργοί και οι πρόεδροι mm. να είναι και αυτοί άμεσα εκλεγόμενοι. Γιατί η υπεμπτουσία της δημοκρατίας είναι να μπορεί κανείς να απολύσει, να διώξει την κυβέρνησή του. Και αυτό είναι πρόβλημα. Κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία είχαμε ένα σύστημα όπου ε, μπορούσε κανείς να εκλέξει την κυβέρνηση και μετά από 4-5 χρόνια να τη διώξει. Αυτό όμως δεν ισχύει πια γιατί η ουσιαστική κυβέρνηση είναι στις Βρυξέλλες, ε, κυβερνούν οι θεσμοί των ε, Βρυξελών. Είτε λοιπόν θα το φτάσουμε μέχρι τέλους ή αν θέλετε θα πρέπει να δεχτούμε ότι θα υπάρχει δυσαρέσκεια από τους πολίτες όπως έγινε στη Μεγάλη Βρετανία που ψήφισαν να φύγουν. Εγώ πιστεύω στη δημοκρατική διαδικασία, πιστεύω ότι οι βουλευτές είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να επιλέγουν την ε, Κομισιόν, ε, θα πρέπει να μπορούν να γίνονται υπουργοί και θα πρέπει να είναι και άμεσα ε, εκλεγόμενος ο πρόεδρος. Θα υπάρχει έτσι λογοδοσία που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι προτάσεις είναι χρήσιμες. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ισηγητά, θα ήθελα πολύ σύντομα να πω ότι όντως εμείς παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο ένα πακέτο, μία έκθεση ε, με πολιτική κατεύθυνση, μία έκθεση ε, και για το 2017 αλλά και για το τι έχουμε καταφέρει τα τελευταία τρία χρόνια στο άρθρο 25 ε, στο οποίο θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ήταν ε, το εργαλείο ηλεκτρονικής εκμάθησης το οποίο αναπτύξαμε για να μπορέσουμε να το διαθέσουμε σε τοπικά γραφεία για να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν ε, τα θέματα της ελεύθερης κυκλοφορίας όπως επίσης και προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες προκειμένου να μειωθούν. Επίσης, Αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προσπαθούμε στην έκθεσή μας να καλύψουμε πολλά σημεία την ε, προώθηση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ιθαγένειας αυτής και τις κοινέ αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσουμε τη συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και την απλοποίηση ε, της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και κυρίως ενίσχυση της προώθησης ε, της ισότητας. Είπατε βεβαίως ε, ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ε, και αυτή είναι μία από τις ε, κύριες προτεραιότητες που είχαμε στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, να υπάρξει ευαισθητοποίηση και σχετική εκστρατεία για την αύξηση της γνώσης των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ηθαγένειας, όπως επίσης και τα δικαιώματα της προξενικής προστασίας ε, και τα εκλογικά δικαιώματα. Στο πλαίσιο της προξενικής προστασίας, ε, που είναι ε, κάτι το οποίο αναφέρεται στην, στο σχέδιο γνωμοδότηση, θέλω να σας αναφέρω μια δημόσια διαβούλευση που έχει σκοπό να δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα, για τα έγγραφα, τα ταξιδιωτικά, τα κατεπήγοντα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει γίνει από την επόμενη εβδομάδα και κάτι ακόμη Επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται όπως για παράδειγμα ε, ενίσχυση ε, της γνώσης. Θα θέλαμε απλώς να σας πούμε ότι υπάρχει ένας κατάλογος Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέσιμος. Ε, θα θέλαμε να σας, βοηθεί, να σας ζητήσουμε να μας βοηθήσετε να εφαρμόσουμε αυτόν τον κατάλογο δραστηριοτήτων που έχουμε προβλέψει στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σόγκορ, έχετε τελικά καταληκτικά σχόλια. Όχι, ευχαριστώ. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Πάμε αρκετά γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο δεν εδώ η εισηγήτρια για το επόμενο ε, θέμα, που είναι οι πτυχέ των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη ένταξη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα άρχισε στις 3.30. Φαντάζομαι ότι θα έρθει η Σοράγια Πόστ ε, στι 3.30. Μέχρι τότε όμως, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Colleagues, if you would like to take your seats again, we can begin. Um, our rapporteur is here. Ήρθε η συγχετριά μας. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, αν μπορείτε να καθίσετε, αν θέλετε βέβαια να συμμετέχετε στη συζήτηση. Παρακαλώ, καθίστε για να αρχίσουμε. Περνάμε στο σημείο 4 που είναι το σημαντικό θέμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και σχετικέ πτυχέ, ένταξη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πολέμηση τη Σωρά η Πόστ είναι η συγκήτριά μα. Ε, η κυρία Πόστ παρουσίασε το σχέδιο έκθεσή τη ε, στην τελευταία μα συνεδρίαση. Όπω θυμάστε, αυτό ήταν πριν από τι καλοκαιρινέ διακοπέ. 252 τροπολογίες έχουν κατατεθεί από τα μέλη της Επιτροπής μας και τώρα θα περάσουμε στην εξέτασή τους. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Σοράγια Πόστ να πάρει το λόγο και να μας παρουσιάσει, να μας πει ορισμένα πράγματα για τις τροπολογίες αυτές πριν δώσω το λόγο στους Κιώδης και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Σοράγια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα. Ε, πραγματικά έχω πολύ μεγάλη όρεξη για το νέο αυτό εξάμεινο ε, που ξεκινάει τώρα, το εξάμεινο εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι πολύ που ξαναβλέπω όλους τους συναδέλφους μου. Ε, χαίρομαι που τόσο πολλοί συνάδελφοι αφοσιώθηκαν στο θέμα και ε, κάναν τον κόπο να καταθέσουν τις τροπολογίες τους, 252 το σύνολο, συνάδελφοι και από την Επιτροπή μας, αλλά και από την Επιτροπή Γυναικών. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες ε, υποβάλλουν πολύ καλές προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αθηγανοφοβίας στην Ευρώπη. Οι περισσότερες δείχνουν ότι, είναι κατανοητό πλέον το γεγονός ότι όταν μιλούμε για το θέμα των Ρωμά δεν θέλουμε να παραγνωρίζουμε το θέμα της, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ε, φτώχειας. Όμως ε, οι βασικές αιτίες των δύο αυτών ε, φαινομένων είναι η αθηγανοφοβία, ε, εκδηλώσεις μίσους, ε, λόγος μίσους κατά τον Ρωμά, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι Ρωμά, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν, μπορούμε, αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, δεν θα υπάρξει βελτίωση στη ζωή των Ρωμά. Όσα προγράμματα και αν υπάρξουν ε, από τα κράτη-μέλη της Ένωσης ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εφαρμοστούν ε, με ε, περιεκτικό και μη διακριτικό τρόπο. Κάποιοι εξημών έχετε υποβάλει τροπολογίες εξίσου ε, καλές ε, νομίζω ε, και με την ίδια κατεύθυνση με τη δική μου, ίσως με πιο ήπια διατύπωση. Ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις κοινωνικές της ευθύνες για, την, τους Ρωμά που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο εδώ και 800 χρόνια. Η κατάστασή τους όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα και πιστεύω ότι εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβουμε μία ισχυρή ε, θέση. Επίσης υπάρχει, υπάρχει μία ε, ριζοσπαστικοποίηση και μία τάση προς το έγκλημα ε, που συνδυάζεται με τους Ρωμά και δεν είναι δυνατόν να γίνεται τέτοιου είδους συλλογική αξιολόγηση μιας ομάδας ανθρώπων. Πολλοί κατηγορούν τους Ρωμά λέγοντας ότι ε, για ποιο λόγο θέλουν ας πούμε, να δουλέψουν και να ε, μορφωθούν. Ποτέ δεν έχω ε, γνωρίσει κανέναν που να θέλει να είναι φτωχός, που θέλει να δει τα παιδιά του χωρίς προοπτικές. Ε, οπότε παρακαλώ ας, ας σκεφτούμε για ένα λεπτό ότι το ίδιο πράγμα θέλει ο κάθε Ρωμά για το παιδί του. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι θα συνεχίσει η καλή μας συνεργασία με τους συναδέλφους ως, ως ε, ε, για, για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ε, η πρώτη μας συνεδρίαση θα γίνει την Πέμπτη και η επόμενη κατά την εβδομάδα του Στρασβούργου και θα γίνει έκθεση, ψηφοφορία της έκθεσης στις 28 Σεπτεμβρίου και θα περάσει στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Σοράγια. Να δώσω τώρα το λόγο στις Κύριε Σόγκορ, θα μιλήσετε εκ μέρους του κύριου Τσάκη. Κύριε Σόγκορ, εκ μέρους του ΕΛΚ, λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Δυστυχώς ο κύριος Τσάκη δεν μπορούσε να είναι εδώ, οπότε μου, διά... μου ζήτησε να διαβάσω την, ε, την δήλωσή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την, το σχέδιο γνωμοδότησής της. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Είναι ε, ότι η αθηγανοφοβία είναι επαρκτό φαινόμενο ε, στις κοινωνίες μας και δημιουργεί ακόμη περισσότερες δυσκολίες ε, στη ζωή των Ρωμά. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, πρέπει να το δούμε από διάφορε οπτικέ γωνίε και ότι, ελπίζω ότι κάποιε από τι προτάσει μου θα βοηθήσουν ε, στην προώθηση ε, της ε, καταπολέμησης της ε, αθηγανοφοβίας. Ε, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο ε, για τα προβλήματα, αλλά και για τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα σε κάποια κράτη-μέλη. Με πολύ χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας, με όλους τους συναδέλφους και ελπίζω μέχρι το τέλος του μήνα να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που είναι αποδεκτό για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σόγκορ. Υπάρχουν κάποιες σκιώδεις που δεν έχουν έρθει. Πάμε στην κυρία ε, Βίλξρομ από τη, Τουσάλντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ο, τους συναδέλφους ε, για όλη την προσπάθειά τους και τις τροπολογίες που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Είναι γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες κοινωνίας των πολιτών. Είναι κείμενο το οποίο πραγματικά έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια μετάβαση ως προς τον τόνο, κάτι το οποίο χρειάζεται ε, στο θέμα της, στη συζήτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για ε, μια ε, μεγάλη ομάδα ανθρώπων που ζουν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης Νομίζω ότι ε, έχει περάσει καιρό από τότε που αρχίσαμε τη συζήτηση με τη Σωράγια για Post. Ε, πάντοτε ήθελε να ε, καταλήξουμε σε ένα πάρα πολύ φιλόδοξο κείμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, παρουσιάσαμε τις περισσότερες τροπολογίες από κοινού και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Γνωρίζουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ένα ζήτημα αριστεράς ή δεξιάς, είναι ένα ζήτημα ανθρώπινο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα στο πλαίσιο του οποίου ε, μπορούμε να δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ των πολιτικών ομάδων και όσον αφορά ε, την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κοινοτήτων Ρωμά της Ευρώπης δεν έχουμε ακόμη αναλάβει πλήρως ε, τις δημοκρατικές ε, ευθύνες μας και πρέπει να πω ότι η κυρία ε, Πόστ πρέπει να χαίρει τη εκτίμηση όλων μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και έχει έρθει επιτέλους ε, η χρονική στιγμή να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ε, βλέπουμε τις κοινότητε Ρωμά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ χαρά θα περιμένω να συνεχίσουμε τον επικοδομητικό μας διάλογο και πρέπει μία ακόμη φορά να τονίσουμε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρξει μία ισχυρή συμμαχία ε, για τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα επιτέλους πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει εμείς ε, στο Κοινοβούλιο να διορθώσουμε όλα τα λάθη που έχουμε διαπράξει στο παρελθόν ε, και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προς τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τη Σοράγια και ευχαριστώ όλους ε, όσους ε, έχουν σκοπό να επενδύσουν χρόνο και κόπο σε αυτό το θέμα. Gracias. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Αλμπιόλα από την ΚΟΕ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Πόστε, για τη γνωμοδότησή της. Εξαιρετική δουλειά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ε, την καταπολέμηση του αθηγανισμού στις πολιτικές τους οριζόντια και θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη δουλειά για την καταπολέμηση αυτής τη συγκεκριμένη μορφής διάκριση, η οποία καταδικάζει στην περιθωριοποίηση και στην ένδυα πάνω από το 50% των αθήγανων τη Ευρώπης. Ε, η συνεργασία με την εισηγήτρια μας επίτρεψε να επιβεβαιώσουμε μια σειρά από τροπολογίες ε, που ε, περιλαμβάνουν μια άποψη του αθηγανισμού ως μια μορφή ρατσισμού και διακρίσεων. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία πτυχή εκτός της έκθεσης αυτής της μορφής διάκρισης. Δεν αναφερόμαστε μόνο στην έλλειψη ένταξης αυτών των ανθρώπων, ε, ε, αλλά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις από τα θεσμικά όργανα ε, υπήρξε και συζήτηση και ρητορία μίσους εδώ, ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, χρειαζόμαστε πολιτικέ κατά των διακρίσεων και του αντιαθηκανισμού που να καλύπτουν όλους τους τομείς. Ε, δεν είναι ε, χρήσιμο να γίνονται δηλώσει καλών προθέσεων τη μία μέρα και ταυτόχρονα να υποστηρίζονται τα πολιτικές ε, περικοπών στον προπολογισμό ή πολιτικέ λιτότητας που ουσιαστικά δεν επιτρέπουν στους δημόσιους οργανισμούς και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις να ε, δραστηριοποιηθούν και ε, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται βαρύγδουπες δηλώσεις όταν ταυτόχρονα έχουμε και ε, προνομιακές σχέσεις με χώρες οι οποίες προωθούν τις διακρίσεις αυτές και ταυτόχρονα να υπάρχει μια μεταναστευτική πολιτική που τα άτομα τα οποία διώκονται επειδή ακριβώ είναι αθήγκανοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία ή εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπλέον, για να ολοκληρώσω κιόλα, ε, θα τονίσουμε και επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δωρεάν δημόσιε υπηρεσίε, ποιότητα όμω δημόσιε υπηρεσίε, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τι ανισότητε σε τομεί όπω για παράδειγμα είναι η παιδεία και η στέγαση. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να αναθεωρήσουμε τι πολιτικέ που εφαρμόζονται μέχρι τούδε, διότι διαπιστώθηκε ότι με κονδύλια τα οποία προορίζονται για την ε, καταπολέμηση του αντιαθηκανισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κατασκευάστηκαν σχολεία τα οποία δεν επιτρέπουν σε Ρωμά να φοιτούν. Ε, αυτές είναι οι πιο σημαντικές τροπολογίες που υποβάλαμε, αλλά βεβαίως θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και στην με τους οργανώσεις στο Ρωμά διότι είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το μίσος με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Μποντήλ Βαλέρο για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Σωράγια για αυτή την πολύ φιλόδοξη ε, δουλειά που έκανε σε αυτή τη γνωμοδότηση και να την ευχαριστήσω διότι θέλεις να ε, συμπεριλάβει όλους εμάς. Ε, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την απόψή μας και να συμπεριληφθούν οι απόψεις μας ευθύ εξ αρχής και θα ήθελα να την ευχαριστήσω τη Σωράγια. Συμφωνώ και εγώ μαζί της, χρειαζόμαστε ε, στεναρές δηλώσεις σε αυτό το κείμενο διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ρωμά είναι πολίτες ε, δεύτερης κατηγορίας ε, στις χώρες μας και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον μια κατάσταση, όπου η ελευθερία ε, μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών αμφισβητείται σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Όχι δική μας ελευθερία κυκλοφορίας ως άτομα που, τα οποία ζουν αλλά η ελευθερία των Ρωμά που έρχονται στις χώρες μας και ε, ζητιανεύουν στους δρόμους. Η δικιά, του ελευθερία, η δικιά τους ελευθερία κυκλοφορίας αμφισβητείται. Αλλά όλοι οι μετανάστες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να την χάνουν τις ίδιες μεταχείρισης. Ε, πολλά συμβαίνουν ε, με τις, ε, στις διάφορες χώρες με τους Ρωμά και αντί να προσπαθήσουμε να διαρευνήσουμε τα αίτια και τους λόγους για τους οποίους έρχονται στη χώρα μας οι Ρωμά και ζητιανεύουν στους δρόμους, αντί να αναζητήσουμε λοιπόν τα αίτια, πολλοί θεωρούν ότι η καλύτερη λύση είναι να απαγορευτεί το φαινόμενο. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να ε, βρούμε τους λόγους για τους οποίους κάποιος είναι διατεθειμένος να φύγει από τη χώρα του, να αφήσει πίσω ε, όλη του την οικογένεια ή τα παιδιά του για να πάει να ζητιανεύει σε μια άλλη χώρα. Δεν νομίζω ότι κανένας θα θέλει να ζητιανεύει σε μια ξένη χώρα αντί να έχει μια θέση απασχόληση σε μια άλλη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχουν και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά παρά το γεγονός ότι υπάρχει και ο χάρτης ε, και υπάρχουν και όλα τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα δικαιώματα ε, που πρέπει να προστατεύουμε, δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι για να τιμωρηθούν οι χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται και δεν ε, ε, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία ώστε να μπορέσουμε με να επιβάλλουμε κυρώσει σε χώρε οι οποίε δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν αναφέραμε μόνο στου Ρωμά, πολλοί άλλοι πλήττονται από αυτή την κατάσταση. Δεν έχουμε όμω αυτή τη στιγμή ε, μεθόδου ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορέσουμε να ασκήσουμε πιέσει σε αυτέ τι χώρε. Δεν αρκεί βεβαίω να υπάρχει απλώ ε, νομοθεσία. πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Και εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε απόψεις και χαίρομαι που μπόρεσα να συμμετέχω σε αυτή την έκθεση και να προσυπογράψω και πολλές από τις τροπολογίες και της Οράγια αλλά και των άλλων συναδέλφων. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα πάρα πολύ καλό και ισχυρό κείμενο εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Ε, προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει στρατηγικό ρόλο σε όλο αυτό το θέμα. Ε, πριν λοιπόν επανέλθουμε στη Σοράγια, ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής του κ. Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρέμβω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για αυτή την πραγματικά θαυμάσια έκθεσή της. Συγχαρητήρια κυρία Πόστ. Είναι μια έκθεση όχι μόνο πολύ καλά δουλεμένη, αλλά είναι και μια έκθεση επί της ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του με στεναρό τρόπο, να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά στην ενσωμάτωση των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει ε, την υποστήριξή τη ε, προς όλες τις τροπολογίε προς το γεγονός ότι υπήρξαν τόσε πολλέ τροπολογίε, περίπου 250 και νομίζω όλες ε, στηρίζουν και τάσσονται υπέρ του μηνύματο που εκφράζει η κυρία Πόστ. Επιτρέψτε μου επίσης να υπογραμμίσω ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το 2011 έχει επεξεργαστεί το πλαίσιο για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Και τώρα έχει έρθει η στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε μετά το 2020. Και όλα αυτά έρχονται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ε, το Κοινοβουλίο τοποθετείται ε, για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Έτσι λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα με όλα αυτά που είπατε. Επίσης, ε, συμφωνούμε με πάρα πολλές ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους ε, σκιώδης ηγητές που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, ίσως μερικές φορές με διαφορετική διατύπωση. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια 800 χρόνια αντιαθηγανισμού με διακρίσεις και μόνο 5-6 χρόνια μιας κοινή ενωσιακής προσπάθειας για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση και στην έκθεση υπάρχει πολύ καλή ισορροπία, επισημαίνονται τα αίτια, αλλά παράλληλα εξετάζεται και η μερίσια διάταξη το όλο θέμα του αντιθέτου Αφιγανισμού να βρούμε μια καλή ισορροπία να είναι ικανοποιητική η ισορροπία αυτή, να είμαστε σκληροί αλλά όχι και αποθαρρυντικοί. Ε, σημειώνουμε πρόοδο, ε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης ε, θα ήθελα να επανέλθω για αυτό το θέμα της ε, ελεύθερης μετακίνησης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι απόλυτα σαφές ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την υποστήριξή μου στις τροπολογίες 124 και 135 της κυρίας Μπίλτ από τη Σουηδία. Αυτές οι δύο τροπολογίες τοποθετούνται πάνω σε αυτά τα δικαιώματα, λένε ότι είναι αδιαπραγμάτευτα και είναι η αρμοδιότητα των κρατών μελών να εκδίδει τις ταυτότητες, επί παραδείγματι. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην προκαλείται η εντύπωση ότι παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα. Και τέλος, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με την κυρία Πόστ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσε να υπάρχει έτσι σε κάποια σημεία μια πιο ήπια διατύπωση. Δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό να γίνεται επισήμανση της, των εγκλημάτων και της εγκληματικότητας ως Ρωμά. Ε, δεν ταιριάζει αυτό. Ίσως είναι θέμα διατύπωσης και ορολογίας, αλλά να δούμε πώς μπορεί να διατυπωθεί αυτό το θέμα. Προσβλέπω λοιπόν στην ε, τελική διατύπωση των τροπολογιών. Ε, ελπίζουμε να είναι συμβαστικές τροπολογίες που θα αποτελούν την ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική ένταξη και τον αντιαθηγανισμό αν έχει κάνει μια τέτοια έκθεση όπως αυτή που έχουμε μπροστά μας, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ε, την, ε, το πλαίσιο πολιτικής ε, μετά το 2020. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσουμε την κυρία Πόστα και τους σκιώδεις εισηγητές που μας επισήμαναν το θέμα αυτό. Νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι οι 252 τροπολογίες διαφέρουν ε, από τη ε, από άλλες τροπολογίε που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν. Τώρα έχουμε πολλά νέα στοιχεία. Στοιχεία ε, που εξετάζει η Επιτροπή μας. Ε, πριν από 20 χρόνια υπήρχαν θέματα διακρίσεων, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές και την εισηγήτρια για την τοποθέτησή τους που φαίνεται μέσα από τις 252 τροπολογίες. Και τώρα θα θέλω να απευθυνθώ στην εισηγήτρια να δώσω το λόγο για τις καταληκτικές της ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Σμίτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση Justice. Ε, ε, είναι δύσκολο να εξευρεθεί ισορροπία γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αθηγανοφοβία. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν. Οπότε είναι σωστό ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Ευχαριστώ λοιπόν και τους κοιόδης εισηγητές και τους ε, υπολείπους συναδέλφους. Νομίζω είναι σημαντικό να είμαστε διαφανείς και να, το, να συνεργαστούμε γιατί όπως είπε και η Σεσίλια, δεν είναι ζήτημα αριστεράς ή δεξιάς, δεν είναι θέμα ε, πολιτικής ε, οικογένειας, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει κανένα ε, χρώμα. Το μόνο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι την ακροδεξιά και τους φασίστες που μερικές φορές κάνουν επιθέσεις, ακόμη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει λοιπόν να λάβουμε την ευθύνη μας ως προς αυτό, γιατί δεν αποδεκτώ ε, το 2017 αλλά και στο μέλλον ε, να είμαστε περήφανοι ως πολιτικοί αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση των 10 εκατομμυρίων περίπου Ρωμά. Εγώ δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ζήσω καλά γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι ε, που ζουν δίπλα στους ε, κάδους απορριμμάτων, ε, νέα παιδιά, που μικρά παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο γιατί δεν έχουν νερό, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν πρόσβαση ε, σε μολύβια και τετράδια ή επειδή υπάρχει διαχωρισμός. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο και νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας και βεβαίως ε, περιμένω ε, με μεγάλη αγωνία τις συζητήσεις με τους σκιώδεις. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που δεν θα χάνει την ουσία της έκθεσης. Από ό,τι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, again to you and the... Ευχαριστώ πολύ. 28 Σεπτεμβρίου έχουμε προγραμματίσει την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Πάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωση Αφρικής, μια όθεση για την ανάπτυξη θα παρουσιαστεί το σχέδιο γνωμοδότησης, ε, επί της ουσίας υπεύθυνη η Επιτροπή Ντέβε, Σεσίλ Κασέτου Κιέγκε, είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησής μας. Μόλι oh, Μόλις ε, με ενημερώνουν ε, ότι ναι μεν η συγγήτρια είναι εδώ, στην ώρα της, αλλά οι σκιώδεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν προσέλθει ακόμη. Ε, σκιώδης ηγετής από το ΕΛΚ είναι εδώ όμως. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε και θα έρθουν και οι υπόλοιποι σιγά σιγά. Εντάξει. Από όσο έλεγα λοιπόν, ε, τον Ιούνιο στις 29 είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕ για μια κοινή ανακοίνωση για την ανανεωμένη στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρικής ε, για το θέμα της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης ε, και σε αυτό το σημείο ακριβώς εστιάζεται η κυρία Κιέγγε. Ε, Στι 12 Ιουλίου είχαμε λοιπόν την πρώτη τελεγή απόψεων και ακούσουμε τώρα την άποψη τη συντάκτρια νομοδότηση και μετά των σκιωδών ε, εισηγητών. Τουλάχιστον είναι εδώ σκιώδη ε, του ΕΛΚ και από ό,τι κατάλαβα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσέλθει και εκείνη σύντομα. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα την άποψη τη εισηγήτρια. Τη δίνω το λόγο. Σε σύλληχη το λόγο. Ευχαριστώ Κλοντ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης επικεντρώνεται στην ε, διαχείριση της μετανάστευσης και της κοινοτικότητας, ε, παράγοντες που είναι καθοριστική σημασία σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας για τη σταθερότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προσπάθειες από κάποιες κυβερνήσεις ε, το τελευταίο καιρό, ο αριθμός των ε, μεταναστών και των ετούντων άσυλων που φτάνουν στην Ευρώπη δεν αλλάζει, δεν θα μειωθεί. Οι διαδρομές αλλάζουν, αλλά ο αριθμός όχι. Εάν δεν λάβουμε υπόψη όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και του μεταναστευτικού φαινομένου, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να περάσουμε από την κοινωνία των πολιτών και τη διασπορά και την τοπική κοινωνία για να μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα βαθύτερα αίτια των μεγάλων μετακινήσεων των προσφύγων και των μεταναστών και να αναγνωρίσουμε και τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ελευθερίες σε ανθρώπους οι οποίοι ξεφεύγουν από πολέμους, από φτώχεια και δίωξη. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής, ε, διέλευσης και προορισμού. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην καταπολέμηση της ε, εμπορίας ανθρώπων και να χρησιμοποιήσουμε και ε, διάφορα άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα χρηματοοικονομικές έρευνες. Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης νόμιμες και ασφαλείς διαδρομές και πρέπει να διευκολύνουμε και την κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων στην Αφρική και μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη και η Αφρική έχουν κοινό συμφέρον και κοινή ευθύνη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου. Εάν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να συνεισφέρουμε και να δώσουμε μια νέα όθηση για την ανάπτυξη, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε ότι αν γίνει κατάλληλη διαχείριση, η κινητικότητα και η μετανάστευση μπορούν να βοηθήσουν να πλουτίσουμε και να ενισχύσουμε τις κοινωνίες μας, να δώσουμε νέα όθηση στην ανάπτυξη, να προωθήσουμε τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, αλλά και την χρηστή διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ και εν αναμονή των σχολείων σας θα μπορέσω στο τέλος να κάνω και μια τελική αξιολόγηση. Ευχαριστώ και θα πρέπει να αναφέρω ότι δεν υπάρχει κανείς ε, πιο ε, άξιος να κάνει αυτή την γνωμοδότηση γιατί κάνεις και εξαιρετική δουλειά στην εταιρική σχέση με την Αφρική. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, εκ μέρου των σχεδόν εισηγητών, εκ μέρους της κυρίας Ντατίν, η κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και όπω είπατε αντικαθιστώ ε, τη Ρασίδα Ντατή η οποία δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Καταρχά, η Ρασίντα θα ήθελα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότηση για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο αποφασίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση να επικεντρωθούμε στι συγκεκριμένε αρμοδιότητε τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η εισηγήτρια αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με το ρόλο των θεμάτων μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή στρατηγική και πραγματικά όντω εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε και επαναλαμβάνουμε ότι εδώ στην Επιτροπή μα δεν θα μπορέσουμε να βρούμε βιώσιμη λύση στην μεταναστευτική κρίση εάν δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και τη Αφρικανική Υπήρου. Η συνεργασία με τι χώρε τη Αφρική θα πρέπει να εδρεωθεί και θα πρέπει να προωθήσουμε την δημιουργία ε, συμφωνιών επανεισδοχή, οι οποίε θα γίνονται και απόλυτα σεβαστέ, ισχυρέ εταιρικέ συμπράξει με χώρε τη Αφρική για να προσφέρουμε μεγαλύτερε ευκαιρίε για του πολίτε και στι δύο επίρους. Ε, κατά την άποψη τη ε, τη λείπει μία πτυχή ακόμα. Θεωρεί ότι η συνεργασία στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτή στη γνωμοδότηση. Η τρομοκρατία δεν είναι απλώ ε, σημαντικό αίτιο τη μετανάστευση, αλλά αποτελεί και πρόσκομα για να δημιουργήσουμε ευημερία και ανάπτυξη και ασφάλεια για τους πολίτες δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι ε, η ειρήνη, η σταθερή δημοκρατία και ευκαιρίες για τους νέους μας ε, είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε, αλλά η τρομοκρατία αποσταθεροποιεί πάρα πολλές χώρες, οι οποίες ήταν ήδη ιδιαίτερα ευάλωτες. Ομάδες όπως η Μπόκο Χαράμ προσπαθούν να καταστρέψουν αυτό το οποίο δημιουργούμε και η τρομοκρατία είναι παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο έχει συνέπειες και για τις δύο υπήρους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε αυτή τη γνωμοδότηση, η σκιώδηση συγγήτριά μας θα ήθελε να ζητήσει μεγαλύτερη συνεργασία συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να μπορέσουμε να πατάξουμε τρομοκρατικά δίκτυα. Θα πρέπει να υπάρξει και καταπολέμηση της χρηματοδότησης τη τρομοκρατίας επίσης. Θα υποβάλει λοιπόν και σχετικές τροπολογίε και προσβλέπει στη μελλοντική συνεργασία με την ε, εισηγήτρια και τους άλλους και όδης ε, ε, στις επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ, Ιμπότιλ Βαλέρο, για τους πρασίνους. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Σεσίλ ε, να προσθέσω μερικά πράγματα. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες ε, μπροστά μας, θα καταθέσουμε τροπολογίες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορούμε την αναπτυξική βοήθεια να την ε, συνδέουμε με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους. Στο σημείο υπαριθμών 3, εκεί γίνεται λόγος για θεομηνίες, αλλά δεν γίνεται καθόλου λόγος για την κλιματική αλλαγή. Οι φυσικές καταστροφές μπορεί να είναι η συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτό δεν είναι και απολύτως απαραίτητο και ισχύει και το αντίθετο. Η κλιματική αλλαγή δεν οδηγεί απαραίτητα σε φυσικές καταστροφές. Μπορεί παραδείγματο χάρη να έχουμε ε, ξηρασία διαρκείας που αναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να ε, μεταναστεύσουν σε μεγάλες πόλεις. Ε, ή αν θέλετε να ταξιδέψουν, να διασχίσουν τη θάλασσα για να μετεγκατασταθούν ε, κάπου αλλού. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, παρουσιάζουμε την ευρύτερη προοπτική και όχι μόνο την κλιματική αλλαγή. Και κάτι άλλο που ενδιαφέρει είναι η ε, νόμιμη με, μετανάστευση. Οι μετανάστες οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, δεν διώκονται, είναι οικονομικοί μετανάστες. Θέλουν να μεταβούν κάπου αλλού για να μπορούν να φροντίσουν την οικογένειά τους. Και αυτούς πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Αυτοί υπάρχουν, έρχονται σε εμά ε, και δεν έρχονται πάντα με νομότυπο τρόπο στην Ευρώπη. Ε, ένα άλλο που πρέπει να δείξουμε είναι τα, ε, οι δυνατότητες που έχουν μετανάστες να κάνουν εμβάσματα στις χώρες προέλευσής τους. Υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν καθεστώς, να μην έχουν ε, ε, ταυτότητα και αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να βάσουν χρήματα στις οικογένειές τους. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε. Τους νέους. Να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτούς. Η Αφρική είναι η μόνη ήπειρος που δεν έχει γυράσκουσα κοινωνία. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάρα πολύ χαμηλός σε, σε πολλές ε, χώρες. Αυτό βέβαια οφείλεται πολλές φορές σε συγκρούσεις, στο AIDS, σε επιδημίες. Υπάρχουν αυτά, όχι όπως παλιά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν ε, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε νεαρή ηλικία. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Αφρική και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η Αφρικανή πολιτική εξάλλου το λένε συνέχεια ότι θα πρέπει να επιληφθούμε των νέων. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το προβάλλουμε περισσότερο στη γνωμοδότησή μας. Ο κύριος Βανότην, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη. Φαντάζομαι θα μιλάτε για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική, έτσι δεν είναι. Απλά να πω και εγώ ότι έρχεστε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά βέβαια είστε και αναπληρωματικός εδώ. Ο εκ μέρου του κ. Τίσσαρσον, ο οποίο είναι ο για αυτή τη γνωμοδότηση και που δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα, ζητά συγγνώμη γι' αυτό. Σε τελική ανάλυση Μιλάμε για γνωμοδότηση, αλλά εγώ είδα λιγάκι την αρχική έκθεση και νομίζω ότι η έκθεση αυτή παρουσιάζει πολλές ελλείψεις. Οφείλουμε να τις εξετάσουμε στην Επιτροπή μας. Κάτι το ελάσσον το Κοινοβούλιο παρουσίασε μία έκθεση για την ε, ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Αφρική ε, για την στήριξη ειρηνευτικών διαδικασιών. Τον Ιούνιο του περασμένου έτους έγιναν αυτά. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό για αυτήν την Επιτροπή να τονιστεί αυτό το στοιχείο. Ε, η έκθεση καταλήγει στο ότι το πρόγραμμα χρηματοδότησης ε, δεν αρκεί. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν όροι έτσι ώστε και η Αφρικανική Ένωση να αυξήσει τη δική της τη συνεισφορά σε επιχειρήσει στήριξης της ειρήνης. Και κάτι άλλο που δεν καλύπτεται κατά τη γνώμη μου είναι αυτό το θέμα των ναρκών κατά προσωπικού και όπως ξέρετε αυτό είναι μία ε, μάστιγα στην Αφρική, επηρεάζει την ασφάλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και από αυτού μία συγκεκριμένη αναφορά. Υπάρχει κάποια αναφορά και ως προς την ε, διαφθορά. Ε, νομίζω γίνεται κάποια προσπάθεια να μιλήσουμε για τη διαφθορά και στις ε, δύο υπήρους. Η έκταση της διαφθοράς στην Ευρώπη, που δεν μπορεί να συγκριθεί με το επίπεδο διαφθοράς που υπάρχει σε πολλές αφρικανικές χώρες. Όχι σε όλες, αλλά σε πολλές εξ αυτών. μιλάμε για λαιλασία του εθνικού πλούτου και αυτό είναι σημαντικός παράγων που οδηγεί στην συνεχιζόμενη φτώχεια και εξαθλίωση που υπάρχει σε αυτή την Ήπειρο. Και κάτι άλλο. Πράγματι αυξάνεται ο πληθυσμός. Έχουμε μάλιστα δημογραφική έκρηξη. Και να μην θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Εκεί κατ' ουσίαν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Το μεγάλο όμως θέμα, τουλάχιστον όσον αφορά την Επιτροπή μας, είναι βεβαίως το θέμα της μετανάστευσης. Γνωρίζω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα, γνωρίζω ότι δίστανται οι απόψεις των συναντέλφων επί του θέματος. Ε, μπορούμε να μιλάμε για ε, τα κίνητρα που οδηγούν ε, στη μετανάστευση, αλλά εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια πιο ρεαλιστική και ουσιαστική στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη μετανάστευση. Αναμφίβολα ο στόχος θα πρέπει να είναι να μειωθούν ουσιαστικά για να μην μπούμε να σταματήσουν πλήρως οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές από την Ευρώπη προς την Ευρώπη. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και Δυστυχώς όμως ε, δεν μοιάζει να γίνεται αναφορά επ' αυτού. Στην αρχική έκθεση βρήκα τα κεφάλαια για τη μετανάστευση και αυτά είναι πάρα πολύ αδύναμα. Κατά την άποψή μας, κατά τη δική μου μάλλον άποψη, δεν αρκεί απλά να ζητά κανείς ε, την ενίσχυση της ε, συνεργασίας με ε, χώρες προέλευσης, διαέλευσης και προορισμού. Χρειαζόμαστε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ε, και πρέπει να πω βέβαια ότι με κατησύχασε λιγάκι το γεγονός ότι ορισμένοι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και ακόμα και η εκπρόσωπο τη, είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήθηκαν στο Παρίσι στις 28 Αυγούστου και κατέληξαν σε κάποιε νέε προτάσει για τα hot spot που πρέπει να αναγερθούν σε κάποιε Αφρικανικέ χώρε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα των μεταναστευτικών ροών, τη ασφάλεια των συνόρων, των σωστών ελέγχων. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι μας μπορούμε βέβαια να γράψουμε εκθέσεις ε, για το πόσο θαυμάσια είναι όλα, ε, το τι κάνουν όλοι, ε, αλλά αυτό δεν μας οδηγεί πουθενά. Κύριε Πρόεδρε, Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι στην Επιτροπή δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου. Εγώ παρόλα αυτά πιστεύω ότι στην έκθεση αυτή υπάρχουν πολλές παραλήψεις ε, ε, και θα πρέπει πραγματικά ε, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτές τις παραλήψεις. Ευχαριστώ πολύ. Κάνατε πολλέ προτάσει. Πριν πάω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριο στόχο τη έκθεση κυρία Κιέγκε είναι η διαχείριση τη μετανάστευση και αυτό είναι ο κεντρικό άξονα και τη ε, γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα. Η πρώτη τελεγή απόψεων έγιναν με την ε, ΕΙΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ή άλλω, αλλά θα σα απαντήσει η Σεσίλ Κιέγκε ε, σε όλα όσα είπατε, στο τέλο βέβαια. Κάποιο ακόμη θέλει να πάρει το λόγο. Θα δώσω πρώτα το λόγο στη συνάδελφο και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Σεπολπία όμω δυστυχώς μιλάει με κάποιον τώρα. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Σίπελ, δεν ήξερα ότι ο κατάλογο μιλητών είχε ήδη κλείσει. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ τα σχόλιά μου για αυτή την πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότηση και το ε, τμήμα, το, την αυθύνη που έχουμε εμεί ω ε, Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι είχαμε μία ευρεία συζήτηση την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με μία από τις χώρες μέλη της Ένωσης και πολλοί ομιλητές από διάφορες πολιτικές ομάδες τόνισαν τη σημασία ότι οι κοινέ τους, το ότι οι μας αξίες, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία είναι στο επίκεντρο, είναι το κύριο στοιχείο της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης και ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε αυτές τις ε, Αξίε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε καλή συνεργασία με, την Ευρω... με τις ε, ε, τρίτες χώρες, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ειρήνη, τη δημοκρατία και το, κρά... κράτος δικαίου και στις τρίτες χώρες, έχοντας στο μυαλό μας, ε, όχι μόνο, αλλά επιπροσθέτως, ότι να μην τα καταφέρουμε και να έχουμε διαφθορά και διάφορες μορφές δικτατορία σε τρίτες χώρες, θα έχει ένα αποτέλεσμα την ε, μετανάστευση την οποία μετά εμείς θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε. Ένα ακόμη ζήτημα ως προς τη μετανάστευση, είναι μια έκθεση της ΔΕΒΕ και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, είναι το θέμα της φτώχειας και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προοπτικές για τον κόσμο στις χώρες αυτές. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις τη ζωή σου, φεύγεις από τη χώρα σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έζησαν σε προηγούμενους αιώνες και πολλοί Ευρωπαίοι. Και τώρα υπάρχουν ε, άνθρωποι που έρχονται από την Αφρικανική ε, Ήπειρο ε, στην Ευρώπη για τον ίδιο λόγο. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα, υπάρχει, θα υπάρχουν ε, συνε, και συνεκτικές πολιτικές. Ένα πράγμα είναι να δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια για τη μία ή την άλλη μορφή ανάπτυξης στις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν προοπτικές και που υπάρχει φτώχεια. Και κάτι άλλο είναι να εξασφαλίζουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την αναπτυξιακή βοήθεια δεν αντισταθμίζεται από άλλες πολιτικές οποίες ε, έχουμε όσον αφορά ε, την εμπορική πολιτική μας, ε, την αλληλεία κλπ. Ελπίζω λοιπόν αυτή η έκθεση να αυξήσει την να ευαισθητοποιήσει γιατί ακόμη και στο πλαίσιο της μετανάστευσης, ε, δεν είναι το μοναδικό πράγμα αυτό που πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να δούμε το σύνολο των πολιτικών ε, τις οποίες ακολουθούμε από κοινού ε, με τις χώρες Αφρικανικής Επίρου και να υπάρξει, το να υπάρξει για να υπάρξει μια αλλαγή ε, πρέπει να προσπαθήσουμε όχι μόνο να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τη βελτίωση της κατάστασης, αλλά και διεθνείς εταίροι να συμμετάσχουν ε, και ε, να δοθεί στις τρίτες χώρες η δυνατότητα να μας πιούν τη δική τους άποψη για το τι πιστεύουν ότι θα βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης. Μαρή Κριστίν, μόλις ήρθες, θέλεις να πάρεις το λόγο, είσαι η για την ΚΟΕ. Ξέρω ότι μόλις ήρθες. Θέλεις να πάρεις το λόγο? Ναι, πολύ σύντομα. Συγγνώμη, Συγγνώμη Σεσίλ, ε, ήμουν στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί θα γίνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη και είχε έρθει ο δικός αποσταλμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ακρόαση στην Επιτροπή μας. Θα θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τη Σεσίλ για ε, τη δουλειά της. Άκουσα το τέλος της παρέμβασης της Βίλκιτ, Η ανησυχία μου σε σχέση με αυτό ε, που είπε, αν και συμφωνώ, ε, ε, πρέπει να υπάρχει μία αμοιβαιότητα και να υπάρχει αίσθηση από τις χώρες οποίες προσπαθούμε να βοηθήσουμε ότι όντως βοηθούνται. Και το λέω αυτό σε σχέση με τους Αφρικανούς εταίρους. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια ε, διαβάθμιση. Ε, δεν είναι το ίδιο πράγμα όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όλων των χωρών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την πραγματική κατάσταση των συγκεκριμένων χωρών και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο την εντύπωση ότι οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν προτεραιότητα, επικρατούν ε, στο πλαίσιο των συζητήσεων ε, στην ανάπτυξη των σχέσεων και των συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας. Εγώ, δεν μου άρεσε αυτός ο όρος, οικονομική συνεργασία με την Αφρική, γιατί υπονοεί κατά κάποιο τρόπο ότι Είμαστε σε ισότιμη βάση. Ε, η αφρικανική κατάσταση με την ε, ευρωπαϊκή ε, δυνατότερη οικονομία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν, δεν λέω δεν πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις, αλλά πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις λαμβανομένων υπόψεων των γεγονότων, της πραγματικότητας. Έχουμε την εντύπωση λοιπόν ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ευρωπαϊκά για να τα αποκαλέσω έτσι, βέβαια τα ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν είναι πάντοτε αυτά τα οποία υπερασπίζονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεών μας. Ε, πρέπει και εκεί λοιπόν να, ληφθούν υπόψη, να ληφθεί υπόψη η πραγματική κατάσταση των διαφόρων ε, χωρών. Έχω ε, σκοπό λοιπόν να καταθέσω τροπολογίω. ναι, ναι, μία συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες είναι βασική πρόκληση για το μέλλον, όμως υπό τον όρο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει το ρόλο που ε, της ε, ανήκει, δηλαδή όχι μόνο να δίνει ε, προτεραιότητες ε, στα νέο απεικιοκρατικά ε, συμφέροντα της, έτσι θα τα αποκαλούσα εγώ, αλλά να σκεφτεί και το μέλλον, το πραγματικό μέλλον και τη βελτίωση του μέλλοντος ε, της Αφρικανικής Υπήρου, γιατί αν συνεχίσουμε να βοηθούμε τον εκφυλισμό της κατάστασης όπως το κάνουμε σήμερα, θα δούμε και άλλες καταστροφές που θα είναι πάρα πολύ βαριές για τις μελλοντικέ γενναίες και εμένα αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνη. Okay, thanks. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, δώσω και πάλι το λόγο στην συντακτήρια της γνωμοδότησης. Ξέρω ότι πρόκειται απλώς για γνωμοδότηση, αλλά διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και όλοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εταιρική σχέση με την Αφρική. Και τώρα οι λεπτομέρειες είναι η μεγάλη πρόκληση για τη συνεργασία αυτή. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής, γιατί ήρθατε κατά τη καθυστερημένη. Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει εκ μέρου της Κομισιόν ιδίω όσον αφορά τι εταιρικέ σχέσεις ε, και τις συμφωνίε για τη μετανάστευση. Σύντομα, γιατί έχουμε και ψηφοφορία εντό ολίγου. Εγώ θα μιλήσω ξανά με τις υπηρεσίες εξωτερικής και μετά οι συνάδελφοι από τις ε, ε, Κομισιόν θα απαντήσουν. Εγώ είμαι αναπληρωτής ε, τμήματάρχης για την Αφρική. Ε, χαιρόμαστε για τη δραστήρια ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία της προετοιμασίας ε, της Συνόδου, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την διακοινοβουλευτική διάσταση αυτής της ε, Συνόδου. Ήδη ε, διαβάσαμε με χαρά το σχέδιο γνωμοδότησης, το σχέδιο έκθεσης μάλλον του κυρίου Πόγκα και τώρα εδώ συζητάμε το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που όπως αναφέρθηκε επικεντρώνεται κυρίως στη μετανάστευση. Το βασικό θέμα της Συνόδου, όπως ε, γνωρίζετε, είναι επένδυση στη νεολαία, αλλά η μετανάστευση είναι και αυτή ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί στη Σύνοδο ε, με θέματα ειρήνης, ασφάλειας ε, και άλλα. Το σχέδιο γνωμοδότησης πολύ σωστά αναφέρει τις θεμελιώδεις αρχές αυτής της εταιρική σύμπραξης στη συζήτηση για τη μετανάστευση, αλληλεγγύη, επιμερισμένη ευθύνη, ε, λογοδοσία και αυτές είναι οι αρχές οι οποίες ε, υπενθυμίζονται και στη διαδικασία της Βαλέτας και στο ε, σχέδιο δράσης της Βαλέτας. Χαιρόμαστε επίσης διότι αναφέρεται και τα στοιχεία τα οποία προωθούν τη μετανάστευση, ε, τις μεγάλες προκλήσεις και επίσης ζητά μεγαλύτερη συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Ε, όπως γνωρίζετε υπάρχουν ε, ε, δραματικές εξελίξεις και χάνονται ανθρώπινες ζωές και φυσικά αναφέρεται και το, ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Αφρική στον τομέα αυτό. Ε, προς το παρόν δεν έχω και πολλές ενστάσεις ε, και δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Να πω ότι είπατε εκπρόσωπος ε, συμμετείχε και σε μια ενεδρίαση που διοργάνωσε ο Πρόεδρος Μακρόν για το θέμα αυτό. Εξακολουθεί να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και στα θέματα τα οποία συζητούμε με την ε, Αφρικανική Ένωση και την Αφρικανική Ήπειρο εν γέννη. Ευχαριστώ πολύ. Από την Κομισιόν είπατε ότι θα μιλήσετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται, βέβαια. Ε, έγινε ανταλλαγή απόψεων τον Ιούνιο. Ωραία, ευχαριστώ. Η Σόφη ε, θέλει το λόγο για το θέμα αυτό. Πολύ σύντομα και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα ή δεν ξέρω εσείς ξεκινήσετε νωρίτερα. Ε, το θέμα της ε, εταιρική σχέσης ε, και η αναπτυξιακή βοήθεια, όλα αυτά ακούγονται πολύ ευχάριστα, όμως υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Παραδείγματο χάρη, τι τελευταίε εβδομάδε βλέπουμε εκθέσει στα μέσα ενημέρωση για πολλά ε, χρήματα που δαπανώνται για το ε, Brigade 48, όπω αποσκαλείται, Κατ' ουσίαν είναι εγκληματική συμμορία τι γίνεται. Αυτοί εμπλέκονται στην πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση. Ε, υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο, ε, αλλά δυστυχώς εκεί δεν μπορεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλάμε για εταιρική σχέση, αλλά ό,τι γίνεται λίγο πιο έξω δεν μπορούμε να το αγγίξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ λιγάκι στους ε, ελέγχους που γίνονται για τα χρήματα που δαπανώνται. Αν ας πούμε δαπανίσουμε εκατομμύριο ευρώ για να διδάξουμε στην ακτοφυλακή της ε, Λιβύης ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, τελικά ε, ποιος ελέγχει εκ των υστέρων τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Γιατί ξέρουμε ότι πολύ λίγοι είναι πρόθυμοι να πάνε για να διδάξουν. Και αυτή η ιστορία με την Brigade 48 πολλοί δεν θέλουν καν να πάνε στον χώρο που βρίσκεται αυτή η συμμορία. Γιατί Πώς χταπανάμε λοιπόν τα χρήματα. Η Ιταλία δίνει δισεκατομμύρια ευρώ στη Λιβύη. Εγώ θα ήθελα να ενημερωθώ τι γίνεται τελικά με όλα αυτά. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμόμαστε ότι ο καλός μας ο φίλος ο κ. Μπελουσκόνη συνήψε μια συμφωνία με τον κύριο Καντάφη και δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και επιτυχημένη. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και κρίμα που είναι λίγοι εδώ παρόντες. Δισεκατομμύρια ευρώ που εκταμιεύονται και δαπανώνται για πράγματα που δεν ξέρουμε. Ε, τι προκύπτει, τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να υπηρετήσουμε τους πολίτες μας ε, με δισεκατομμύρια ευρώ από το να τα στέλνουμε στο πουθενά, στην έρημο της Λιβύης. Ε, δεν είναι εδώ πολλοί για να ακούσουν, αλλά το κοινοβούλιο, στο κοινοβούλιο υπάρχουν πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα θέματα. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μπορεί αυτό να είναι μόνο γνωμοδότηση, αλλά πριν περάσω στην εισηγητία να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια διαδικασία και πραγματικά έχουμε θυμώσει λιγάκι. Ε, σχετικά με τη διαδικασία που τρέχει για το Μαλί, το Αφγανιστάν, το Κοινοβούλιο ε, ή αν θέλετε οι δικοί μας οι όροι έχουν αγνοηθεί και θέλω αυτό να καταγραφεί γιατί εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε και θέλουμε γιατί ε, συμφωνούμε σε κάποιο βαθμό με αυτά που είπε ο κύριος Βανόρντο δηλαδή έχουμε διάφορες απόψεις και θέλουμε οι απόψεις αυτές να εισακούνται. Ευχαριστούμε κυρία Ιντενφέλτ που μας υπενθυμίσατε όλα αυτά που δεν εισακούνται και στη γνωμοδότηση και αλλού. Δεύτερον, θέλω και πάλι να υπενθυμίσω στους συναντέλφους ότι η έκθεση αυτή ασχολείται με τη μετανάστευση, την κοινωτικότητα, τις εταιρικέ σχέσεις. Εφημισμός είναι όλα αυτά. Η πραγματική ανάγκη είναι οι λεπτομέρειες. Ε, και νομίζω ε, τώρα όσον αφορά στις λεπτομέρειες ε, θα πρέπει να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Η έκθεση της εισηγήτρια της κυρίας Κιάνγκε είναι πολύ χρήσιμη γιατί η κυρία Κιάνγκε έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με την Αφρική. Θέλει να δουλέψει με αυτή τη γνωμοδότηση. Ε, οι τροπολογίες θα μπορούν να κατευθούν μέχρι την Παρασκευή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο πια στη διάθεσή μας, αλλά θα θέλουμε, θέλουμε να δούμε ε, πώς θα εξελιχθεί τελικά αυτό το θέμα. Γιατί με την Υπηρεσία εξωτερική δράση και την Επιτροπή υποτίθεται ότι πρέπει να προχωράμε γρήγορα και ε, δεν είδαμε να υπάρχει ταχεία πρόοδος. Σας τα λέω όλα αυτά για να σας ε, εξηγήσω ότι για μας το όλο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ε, Σεσίλ, αν θέλεις ε, να απαντήσει σε κάποια συγκεκριμένα θέματα, αλλά και να μας δώσει έτσι και μία γεύση ή πρόγευση του πώς θα είναι η έκθεσή σου, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Κλόντα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για όλα αυτά που μας ε, είπαν και πάρα πολλές από αυτές τις απόψεις θα τις συμπεριλάβω στην έκθεσή μου γιατί ήταν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ε, νομίζω ότι ε, μπορούν πραγματικά να δώσουν μια όθηση στη δουλειά που κάνουμε. Άκουσα να γίνεται λόγος για ρεαλιστική προσέγγιση και ξεκινάω με αυτό. Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς να μπλοκάρει ένα φαινόμενο το οποίο είναι δομικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Η μόνη ε, ρεαλιστική προσέγγιση είναι η ολιστική. Και νομίζω εδώ στην Επιτροπή μας μιλήσαμε διαμακρών για το θέμα αυτό και έχουμε μάλιστα συντάξει και ε, ψήφισμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται πλέον κατανοητό ότι μια ολιστική προσέγγιση, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση για να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό φαινόμενο. Ω Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, όπως ελέγχθη, το να αρχίσουμε να μιλάμε για την τρομοκρατία που βεβαίω έχει συμπεριληφθεί στο σημείο ε, παρτιμοντία ή εν πάση ε, σε κάποιο άλλο θέμα αυτό είναι παραπλανητικό. Πρέπει να έχουμε, όπως σας είπα, μια ολιστική προσέγγιση και όχι να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα θέματα. Και όχι σίγουρα στην τρομοκρατία, γιατί αυτό θα μας απομακρύνει από το στόχο της ε, γνωμοδότησης. Εξάλλου, πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε κάποια στοιχεία, πολλά έχουν λεχθεί και από την Birgit. Ε, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η Birgit. Η δική μου προσέγγιση θα είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή ε, να παραμείνω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα και να μην ε, προχωρήσω, να μην ξεφύγω από μια ολιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 28 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ για την ε, λεπτομερή συζήτηση για ε, τη γνωμοδότηση αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας ως προς την ουσία της. Ε, λοιπόν, στις 5 παρα 20 έχουμε προγραμματίσει την ψηφοφορία, οπότε θα διακόψουμε ως τότε. Παρακαλώ πάρα πολύ όμως να είστε ακριβώς την ώρα σας ε, εδώ για να ψηφίσουμε. Και παρακαλώ να έχετε έτοιμες και τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι, θα αρχίσουμε 5 παρα 20 ακριβώς. colleagues, if everyone is ready, we will... Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Πρόκειται για το σχέδιο εκτελεστική απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της ακριλοφεντανίλης σε μέτρα ελέγχου. Ο Μπρίς Οχτεφέ είναι ο εισηγητή. Αν δεν θέλει να πάρει το λόγο, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Είναι ε, μια ε, ψηφοφορία και μοναδική έναρξη ψηφοφορίας. Just indicate with your hand. Με το χέρι σας. Με το χέρι σας δείξτε. Ναι, έτσι. Lopez Aguilar will be counted. The vote is now closed. Πέρας ψηφοφορίας. 32 ψήφοι υπέρ, ε, μία αποχή, κανένας κατά. Συγχαρητήρια κύριε Ορτεφέ. Τέλος της ψηφοφορίας. Διακόπτουμε μέχρι τις παρατέταρτο και μετά πάμε στο αριθμό 7 σημείο της διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Διακόπτουμε λοιπόν μέχρι τις παρατέταρτο. Αλλά παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα γιατί έχουμε την ανταλλαγή απόψεων πολύ σύντομα. Παρακαλώ μη φύγετε λοιπόν για το τελευταίο σημείο της διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσία σας εδώ σήμερα το απόγευμα. Η απόψινή συζήτηση ολοκληρώνεται με ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε εδώ τον Επίτροπο, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που είναι εδώ και έχουμε επίσης και τον κύριο Γκάρκοφ, ε, διευθυντή του Ιουλίσα. Ε, καλώς ορίσατε κι εσείς. Ε, ε Κύριε Επίτροπε, όσον αφορά την ε, πρόοδο και προς τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, διότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ λοιπόν Δημήτρη που είσαι εδώ σήμερα και θα σας μιλήσει για το θέμα αυτό ε, σήμερα το απόγευμα. Εισαγωγικά να σας πω ότι το σημείο αυτό έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ισχυρότερα και πιο έξυπνα συστήματα πληροφοριών που έγινε πέρσι και φυσικά η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ασχολείται με τα συστήματα πληροφορικής και έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά επανειλημμένως. Έχουμε μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις ε, στον τομέα αυτό βέβαια το σύστημα εισόδου αξίδου, εξόδου, το ETIAS ε, κλπ. Αλλά θα συζητήσαμε και το μελλοντικό τοπίο των συστημάτων πληροφοριών και ε, την ομάδα υψηλού επίπεδου για τη διαλειτουργικότητα και τα συστήματα πληροφορικής. Όπως λοιπόν ε, σας είπα, είναι πολύ σημαντικό να μας μιλήσει ο Επίτροπος για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και φυσικά υπάρχουν πολύ σημαντικά και τεχνικά ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά φυσικά υπάρχει και πολιτική σημασία για τα θέματα αυτά. Ε, καταρχάς λοιπόν να καλωσορίσω τον Δημήτρη που είναι εδώ για να μιλήσει ε, για τα θέματα αυτά και να μας ενημερώσει και από εκεί και πέρα θα δώσω το λόγο στο διευθυντή του Ιουλίσα για να μας ε, πει και αυτός ε, την απόψή του. Ε, χαίρομαι όμως που είναι εδώ ο Επίτροπος και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που μπήκαν στον κόπο να έρθουν εδώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό Δευτέρα απόγευμα. Δήμητρη, έχεις το λόγο λοιπόν για να μας ενημερώσει για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Και να σας καλωσορίσω και μετά τις θερινές διακοπές. Να καλωσορίσω όλους, λέει ο Επίτροπος. Ελπίζω να περάσετε καλά στις διακοπές. Όλοι χρειαζόμασταν ένα μικρό διάλειμμα ε, για τους επόμενους μήνες, διότι δεν θα είναι εύκολοι, αλλά είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και εσάς, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση και πολύ ευχαρίστως να ξεκινήσουμε ε, τη νέα ε, χρονιά εργασιών με αυτή τη συζήτηση. Η εργασία για τις πολιτικές μας συνεχίζεται και νομίζω ότι θα πρέπει να συναντηθούμε αρκετά στο μέλλον. Σήμερα όμως έχουμε αφιερώσει τη συζήτηση στις πιο πρόσφατες εξελίξεις ε, για τη διαλειτουργικότητα και την πρότασή μας να ενισχύσουμε το ίδιο e λύσα που έχει στενή σχέση με αυτό. Δεν θα χρειαστεί βέβαια να σας παναλάβω πόσο σημαντική είναι η ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αρχές επιβολής του νόμου και δικαστικές αρχές, καθώς επίσης και υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις ασφαλείας ε, ε, σήμερα και ε, στο μέλλον και φυσικά να σταθούμε και στο ύψος των προσδοκιών των πολιτών μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ε, αποδείξουν αυτή την εμπιστοσύνη. Εάν δεν ε, ε, υπάρξει μεγάλη δέσμευση, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική και ισχυρότερη ένωση σε θέματα ασφαλείας. Οι επιθέσεις στο Τούρκου, στο Λονδίνο, στη Στοκχόλμη, στο Βερολίνο νωρίτερα αποδεικνύουν χωρίς καμία αμφιβολία ότι η επιθέσεις αυτές ε, θα μπορούσαν να είχαν ε, αποφευχθεί ή θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει ζωή, ζωές αν υπήρχε πιο έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρότερα συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών, ε, στις, οι οποίε θα είναι στη διάθεση των αρχών ασφαλεία, των τελωνιακών αρχών. Χρειαζόμαστε λοιπόν το SIS, το σύστημα πληροφοριών Schengen, το σύστημα VIS, το ETIAS και άλλα. Επίσης, εφαρμόζουμε ταχύτατα και το σύστημα του Ευρωπαϊκού PNR, τον, ε, του Συστήματος Ανταλλαγής ε, Πληροφοριών των Ταξιδιωτών. Το γνωρίζετε αυτό και έχω ζητήσει από τα κράτη-μέλη επανειλημμένως να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων. Εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και μέσω χρηματοδότησης και εμπειρογνωμοσύνης αλλά και με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Στη διάρκεια του περασμένου έτους, ε, λόγω κυρίως ε, των ε, σκληρών μαθημάτων που μάθαμε με τις τρομοκρατικές επιθέσεις, υπήρξε βαθμιδόν αύξηση της χρήσης αυτών των συστημάτων. Το SIS χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ιδιαιτέρως, αλλά πρέπει να γίνουν και πολύ περισσότερα. Και όταν λέω περισσότερα, δεν αναφέρομαι μόνο σε περισσότερα όσον αφορά ποσότητα, δεν ε, θέλουμε απλώς ε, να αυξηθούν τα συστήματα ασφαλείας, υπάρχουν αρκετά συστήματα. Θέλουμε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα συστήματα που έχουμε στη διάθεσή μας και να ε, συμπληρώσουμε τα κενά που διαπιστώνουμε στην αρχιτεκτονική πληροφορική στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ακριβώς προτείναμε μια δέσμη προτάσεων για να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν τον περασμένο Σεπτέμβριο και Ξέρω ότι τα όσα έκανε ο κύριος Κοέλιο για το θέμα αυτό προχωρούν. Προτείναμε επίσης και ένα νέο σύστημα εισόδου-εξόδου, το οποίο θα εξυγχρονίσει πλήρως ε, τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντίαθ Μέρα και την ε, ομάδα των σχεδόν εισηγητών για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο και προσβλέπω και στην τελική έγκριση του κειμένου τον Οκτώβριο. Προτείναμε το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξιδιωτικών Πληροφοριών και Έγκρισης, το ETIAS, το οποίο θα μας επιτρέψει να γίνεται εκ των προτέρων έλεγχος των ε, αιτήσεων ε, θεωρήσεων διαβατηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο ε, του μοσαϊκού, διότι αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε τέτοιε πληροφορίε. Ξέρω ότι η κυρία Γκάλ αλλά και εσείς όλοι ε, εργάζεστε εντατικά επί του θέματο αυτού και γι' αυτό και ακριβώς σας προτρέπω να προχωρήσετε την έγκρισή του το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, τον περασμένο Ιούνιο προτείναμε τη βελτίωση ε, του ε, συστήματος ε, ποινικού μητρώου για τους υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι δικαστές να έχουν ένα πιο ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η συνύπαρξη των κείμενων και προτινόμενων συστημάτων δυστυχώς δεν αρκεί. Τι χρησιμότητα έχουν όλα αυτά τα συστήματα εάν είναι απλώς απομονωμένα και δεν ε, ε, συνεργάζονται μεταξύ των. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαλειτουργικότητα στις πληροφορίες μας για να μπορούν να είναι και εύχριστες. Πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε κάπως τα συστήματα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αρχές επιβολής του νόμου, οι συνοριοφύλακες, οι υπηρεσίες πληροφοριών, όλοι χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες από όλα τα συστήματα πληροφοριών, προκειμένου να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις στην κατάλληλη στιγμή. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει επίσης ε, να ε, δει ε, και τα θέματα της περιορισμένης πρόσβασης σε αρχές επιβολής του νόμου, σε συστήματα τα οποία δεν αφορούν επιβολή του νόμου. Αυτό το κενό αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει πρόληψη, έρευνα, αποτροπή αλλά και δίωξη ποινικών αδικημάτων. Τα νέα συστήματα αιτιάς ε, χρειάζονται διαλειτουργικότητα για να μπορέσουν να συνεπάρξουν με το σύστημα εισόδου-εξόδου, με το SIS και το VIS, το Eurodac και τα στοιχεία της Europol, όπως έχουμε προτείνει. Στη διάρκεια του 2016, η ομάδα εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε εξέτασε τα θέματα αυτά και τις διάφορες αναλλακτικές λύσεις διαλειτουργικότητας. Εξέτασε τα υφιστάμενα αλλά και τα μελλοντικά συστήματα ε, τις βάσεις δεδομένων της Europol και της Interpol, το PRUM και άλλα συστήματα πληροφοριών, προκειμένου να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα κενά στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και επιβεβαίωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση για τη διαχείριση των δεδομένων, για τα σύνορα και την ασφάλεια, όπου όλες οι, τα σχετικά κεντρικά συστήματα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαλειτουργικά. Επιβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα σεβόμενοι πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίω ε, τα θέματα προστασίας δεδομένων. Και αυτό είναι κάτι ουσιαστικό. Ε, επισημάναμε λοιπόν ότι τα διάφορα συστήματα μεμονωμένα θα πρέπει να σέβονται τις ε, αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Θα πρέπει να τηρήσουν τις δικές τους διατάξεις προστασίας δεδομένων και να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία κανόνες ε, για περιορισμό του ε, στόχου τους, ε, ελαχιστοποίηση των δεδομένων και συγκεκριμένους κανόνες για τη διατήρηση των δεδομένων. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεγάλου αδελφού εδώ. Η διαλειτουργικότητα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται ε, κάτι το οποίο έχετε να ε, δημιουργήσει προβλήματα στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ίσα ίσα που θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματά μας ε, στην ασφάλεια, ε, στην προστασία και στην κινητικότητα. Είναι η ευκαιρία μας να προσφέρουμε περισσότερη εύρωστη και έγκαιρη προστασία με πολύ πιο σύγχρονα συστήματα για τη διαχείριση των πληροφοριών μας. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ε, συνεχίσουν να υφίστανται όταν θα υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων αυτών. Γι' αυτό και ακριβώς ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο Ευρωπαϊο Επόπτη ε, Προστασία Δεδομένων συμμετέχουν στενά στην όλη διαδικασία. Έχουν ήδη ξεκινήσει τεχνικές συζητήσει και μαζί σα και με το Συμβούλιο για να υπάρξει μια κοινή συνεννόηση για τα απαραίτητα βήματα για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών μας μέχρι το 2020. Είμαι βέβαιος ότι ε, μέχρι το τέλος του έτους θα μπορέσουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση επιτάπητος για να υπάρξει και διαλειτουργικότητα των ε, συστημάτων πληροφοριών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάρκο και την ομάδα του στο Ιουλίσα e για την ε, συμβολή τους ε, σε αυτό το έργο και όχι μόνο για τα όσα έχουν κάνει ε, ε, για το θέμα αυτό, αλλά και για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Το Ίγιου Λίσα θα είναι ο ακρογωνία λίθος της δουλειάς μας για τη διαλειτουργικότητα και ο οργανισμός ήδη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, ε συνύπαρξη των συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα συστήματα SIS και VAS καθώς επίσης και τα μελλοντικά συστήματα, όπως για παράδειγμα το σύστημα εισόδου-εξόδου και το ETIAS μόλις ε, θα εγκριθούν. Γι' αυτό και ακριβώς και τον Ιούνιο παρουσιάσαμε μία πρόταση για αναφερομένη ε, εντολή του οργανισμού. Η πρόταση αντανακλά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο οργανισμός για να διασφαλίσει ποιότητα ε, δεδομένων και επίσης ε, ο οργανισμός θα φιλοξενεί τα νέα συστήματα πληροφοριών που ανέφερα με τους απαραίτητους φυσικά πόρους προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτά τα νέα καθήκοντα για τη διαλειτουργικότητα. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, προκειμένου να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια των πολιτών μας, θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη των συστημάτων πληροφοριών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συνοριοφύλακες και οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν τα απαραίτητα ε, στη διάθεσή τους, τις κατάλληλες πληροφορίες, την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό ακριβώ είμαι βέβαιος ότι η νέα εντολή της Υγιού Λίσα θα συνεισφέρει προς αυτό το στόχο και φυσικά προσβλέπω και στη συνεργασία μαζί σας για αυτή την ε, πρόταση όπως και για τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, κύριε Επίτροπε και θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Κύριο Γκάκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, λέω εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γκάρκο, Κάρκοφ. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή ε, συζητάμε για μια αλλαγή που γίνεται. Από τη μια Όσα λαμβάνουν χώρα τώρα εξαρτώνται πλήρως από την ανταλλαγή πληροφοριών και από την άλλη υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα στην εσωτερική ασφάλεια, την διαχείριση των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν θα πρέπει ε, πλέον να υπάρξουν άλλα συστήματα. Ε, με αυτή την έννοια η ομάδα εμπειρογνωμόνων είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν ε, σημαντικά ωφέλη από τη διαλειτουργικότητα η οποία φέρνει και πάρα πολλές ευκαιρίες ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ε, κείμενων και των μελλοντικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διαχείριση ε, των σιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι η διαλειτουργικότητα από μόνη της δεν είναι απειλή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε άλλο, η διαλειτουργικότητα προσφέρει ε, ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στη διελειτουργικότητα δεν πρόκειται για την συγχώνευση τραπεζών δεδομένων. Ούτε και όλοι θα έχουν πρόσβαση στα διάφορα συστήματα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα, η αποτελεσματική χρήση των συγκεντρωνόμενων πληροφοριών. Με αυτή λοιπόν την έννοια οι φορές η Γιουλίζα μετά από τα συμπεράσματα της ε, τελικής έκθεσης ε, ε, η Γιουλίζα προσπάθησε να εξετάσει περαιτέρω τα πορίσματα και να προτείνει τη βέλτιστη δυνατή τεχνική λύση έτσι ώστε η διαλειτουργικότητα να γίνει πραγματικότητα. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω έχουμε μία μελέτη των ε, βιομετρικών δεδομένων και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 27 Ιουλίου και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουμε τη δεύτερη φάση για να εξετάσουμε ε, περαιτέρω τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Η μελέτη προτείνει ένα μια δομή που θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για τη χρήση βιομετρικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλήρη συμμόρφωση των κανονισμών για την προστασία των δεδομένων. Ε, υπάρχει και μια άλλη μελέτη, τελειώνει τώρα για τα δεδομένα και αυτή θα προτείνει έναν αποτελεσματικό ευέλικτο τρόπο έτσι ώστε να, ε, να συντάσσονται εκθέσεις ε, ε, που χρησιμοποιούν δεδομένα, το EU Portal. Και αυτό προχωράει, τέλος του μήνα θα έχουμε το τέλος της πρώτης φάσης. Εκεί προτείνεται να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί και κατά τους αμέσως επόμενους μήνες μετά την ολοκλήρωση της ε, φάσης. Εξάλλου και άλλη μια μελέτη έχει ανατεθεί από την Επιτροπή στηρίζεται από την Ιγιου και προβλέπεται ότι το Δεκέμβρη θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την εφαρμογή όλων αυτών των ε, σχεδίων στο μέλλον. Πολύ δύσκολη λοιπόν η δουλειά που έχει γίνει για την προστασία των δεδομένων που αφορά στα κρατημέλη και την EU και για να ολοκληρώσω, η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια και τη διαχείριση των ε, συνόρων στην Ευρώπη. Η γνώμη της Ιουλίζα είναι ότι θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο ε, και γι' αυτό και εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις νέες μας ευθύνες, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στον τομέα της ε, διαλειτουργικότητας και της ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάρκοφ. Συνάδελφοι, θα δώσω τώρα το λόγο σε εσά, δύο-τρία λεπτά. Ε, ο καθένας. Ε, έχετε πολύ ζητήσει το λόγο και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα γίνει έτσι μια πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Σα ευχαριστώ που είστε εδώ. Με, Μετσόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν ήρθα ε, στην αρχή της συζήτησης, αλλά είχαμε μια επίγουσα ψηφοφορία σε άλλη επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τον Διευθυντή και τον Επίτροπο για την παρουσίασή σας και τις προσπάθειες ε, υπέρ της διαλειτουργικότητας των ε, συστημάτων πληροφορητής, όπως γνωρίζετε. Εμεί όχι μόνο το υποστηρίζουμε, αλλά θεωρούμε ότι η βελτίωση τη διαλειτουργικότητας των συστημάτων είναι μία από τι προτεραιότητε τη, ε, ε, κυρίω προ την πρόληψη επιθέσεων στην Ευρώπη. Έχουμε ήδη βάσεις δεδομένων ε, και τα συστήματα τα οποία διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή πρέπει να συνδέονται καλύτερα, ώστε οι συνοριοφύλακε, οι ιδιοκτικέ αρχέ, οι τελωνιακοί, οι υπεύθυνοι για τη μετανάστευση πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στι απαραίτητε πληροφορίε. Αυτό θα οδηγήσει στην ανείχνωση τη χρήση για την ε, καταχώρηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων ε, υπόπτων ε, τρομοκρατών. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι οι σχετικές πολιτικές διατάξεις στο σύστημα εισόδου-εξόδου είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που είπατε προς το τέλος, να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για το επίπεδο ικανοποίησή σας με την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Θεωρείτε ότι πηγαίνουμε αρκετά γρήγορα και αν όχι, όχι πιστεύετε ότι μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, γιατί ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων ε, είναι πολύ σημαντικός και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει πολλές φορές ε, τονίσει όπως και εσείς. Χαίρομαι ιδιαίτερως, πρέπει οπωσδήποτε να προοδεύσουμε γιατί οι πολίτες μας αυτό περιμένουν από μας. Ευχαριστώ πολύ Ρομπέρτα, η κυρία Σίπελ. Πύρκητα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχά να επαναλάβω με πιο απλά λόγια ότι κατάλαβα καλά για το τι μιλάμε. Σήμερα η κατάσταση είναι η εξή. Αστυνομικοί που ψάχνουν ειδικέ πληροφορίε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ανοίγει μια βάση δεδομένων, ε, κοιτάζει τι πληροφορίε που έχει το δικαίωμα να δει, μετακλίνει την βάση δεδομένων, ανοίγει μια άλλη βάση δεδομένων, αναζητά τι πληροφορίε οι οποίε έχει πρόσβαση εκεί, ξανακλίνει τη βάση δεδομένων, ανοίγει μια τρίτη βάση δεδομένων και ούτω καθεξής. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν ε, Σκοπό έχει να αποφύγει αυτό το περίπλοκο σύστημα συλλογή πληροφοριών από διάφορε βάσει δεδομένων. Ε, με ένα κλικ λοιπόν το σύστημα αυτομάτω θα συλλέξει όλα τα δεδομένα τα οποία, ε, στα οποία έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένο αστυνομικό. Καλό ακούγεται αυτό και αν έχουμε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την ε, προστασία των δεδομένων, ακόμη καλύτερα. Όμως η διαλειτουργικότητα δεν ε, υπάρχει έτσι ξαφνικά. Προέκυψε από τα συστήματα που έχουμε, τις βάσεις δεδομένων που έχουμε. Και εντύπωσή μου είναι ότι πριν αρχίσουμε με τέτοιου είδους διαλειτουργικότητα, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε, ε, τις, να πλουτίσουμε περισσότερο, να πλουτίσουμε περισσότερο τις βάσεις δεδομένων και να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη πρόσβαση πρόσβαση στις ε, βάσεις αυτές δεδομένων ώστε να ε, μπορούν να έχουν περισσότερη πρόσβαση και να μπορούν να συλλέξουν και περισσότερες πληροφορίες. Έχω κάποια ερώτηση. Ε, μερικές φορές ε, λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα στο πλαίσιο μιας βάσης δεδομένων γιατί διαφορετικά υπάρχει ένα κενό. Πότε, πώς αποφασίζουμε όμως κατά πόσο υπάρχει ένα κενό, ένα παραθυράκι, αν δεν χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά αυτά που ήδη υπάρχουν στη διάθεσή μας. Η αξιολόγηση λοιπόν των υπαρχόντων μέτρων και της χρήσης τους νομίζω ότι ε, δεν ε, έχει ε, γίνει και τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι θέλουμε να αυξήσουμε την ποσότητα των δεδομένων και δεν μας απασχολεί το κατά πόσο ε, δεν χρησιμοποιούμε τα πολύτιμα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Μιλήσατε και για το PNR. Θα θέλω να επενθυμίσω ότι υπάρχει μία δήλωση από το δικαστήριο γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι συγκεκριμένα ε, το να αναφερθούμε ε, στο PNR Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή και έχουμε τώρα μία δήλωση του δικαστηρίου και αν δούμε το PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, νομίζω ότι υπάρχουν ε, πολύ παρόμοιες ε, ε, ε, πολύ παρόμοια φαινόμενα. Καλύτερα είναι λοιπόν και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση να μην βιαστούμε, να μην σπεύσουμε για αυτό το PNR. Ε, πρέπει να τα ξαναδούμε αν υπάρχουν κάποια κοινά σημεία με το PNR Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά γιατί δεν θέλουμε μετά να έρθει να μα πει κάποιο ότι δεν κάνουμε τα σωστά. Νομίζω ότι καλή, το καλό νομοθετήν συμπεριλαμβάνει και τέτοιου είδου ελέγχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ που τη τηρήσατε το χρόνο σας, για την ώρα τον έχετε τηρήσει όλοι και έχουμε και πολλούς ομιλητές. Σοφή Ινιτφέλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς ε, να πω ποια είναι η δική μου άποψη. Εγώ είμαι υπέρμαχος, μεγάλη υπέρμαχος ε, της ανταλλαγής ε, πληροφοριών μέσω της λειτουργικότητας, υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών ήθελα εγώ, την οποία απέρριψαν τα κράτη-μέλη και το ΕΛΚ. Κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους παρουσιάσεις, σαν αυτές που άκουσα, μου θυμίζει λίγο αυτό τις δηλώσεις πωλήσεων, ότι ε, πώς ε, κάποιο προϊόν μπορεί να σας εξασφαλίσει ένα υπέροχο σώμα, όμως δυστυχώς είναι λιγότερο ε, συναρπαστική η πραγματικότητα. πρέπει να δούμε λοιπόν τις ευκαιρίες μας, αλλά πρέπει να δούμε και τις απειλές και τις δυνατότητες που έχουμε. Να δούμε και το θέμα της διαφάνειας όμως. Γιατί το θέμα είναι το εξή. Κάθε φορά που μας ζητάτε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσουμε ε, με, τα, ε, με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κάνουμε, αλλά όταν θέλουμε μετά να κάνουμε έναν έλεγχο και να αξιολογήσουμε, μας κλείνετε την πόρτα. Αν μας πείτε, ας πούμε, για το PNR, ε, είχατε πει ότι θα χρηματοδοτήσετε με 310 εκατομμύρια ευρώ τα εθνικά συστήματα PNR. Εντάξει, να το δεχτώ αυτό, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν ε, ρωτούσα, αν ε, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις, ε, τα έντυπα αξιολόγηση με τα οποία ζητήσαμε τη χρηματοδότηση και μας είπε όχι. Υπάρχει κακοδιαχείριση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είπε και το δικαστήριο. Μην έρχεστε λοιπόν να μας ζητάτε να σας υποστηρίξουμε και να σας βοηθήσουμε αν δεν μας δίνετε μετά τη δυνατότητα να κάνουμε μία χρήσιμη εποπτεία. Ε, γιατί ε, μας λέτε ότι αυτό θα συνάδει πλήρως με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και ότι θα διαβουλευθείτε με το EDPS κλπ. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, όλα πολύ ωραία, αλλά είμαι αρκετό καιρό εδώ για να ξέρω ότι συνήθως όντως κάνετε διαβούλευση και μετά παραγνωρίζετε ολοσχερός την άποψη του EDPS. Οπότε δεν θέλω να μου πείτε ότι θα κάνετε διαβούλευση, θέλω να μου πείτε ότι θα ακολουθήσετε τις συστάσεις τους. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί όπως είπα Πραγματικά είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια της ανταλλαγής απόψεων, αλλά οι δικλείδες ασφαλείας για τους πολίτες, σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην κάτω χώρες βρήκαμε αυτή τη βδομάδα ότι φορολογικέ φορολογικές αρχές παρανόμως και εσκεμμένως αποθήκευαν εκατομμύρια πινακίδες αυτοκινήτων ε, και μάλιστα ε, ε, μη ακριβή, ανακριβή στοιχεία ε, πολιτών. Αν λοιπόν οι πολίτες υποφέρουν λόγω ε, δεδομένων ανακριβών και που παρανόμως έχουν αποθηκευτεί, αυτά θα τα ανταλλάξουμε με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φαντάζεστε τι θα γίνει. Εγώ συμφωνώ απολύτως λοιπόν με την ανταλλαγή απόψεων, αλλά έχω επανειλημμένος πει ότι πρέπει να υπάρχει μία να, να συμπληρώνονται, να συνοδεύονται από την κλίδα ασφαλείας. Θα ήθελα να ακούσω λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σόλμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ καταρχάς που είστε εδώ κύριε Επίτροπε και μα ενημερώνετε για αυτή τη δουλειά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, να ε, γίνει κατάλληλη ανταλλαγή. Ε, είναι κάτι για το οποίο έχουμε συμφωνήσει και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας. Θα πρέπει να επιτρέψουμε από νομικής, από πολιτικής και από τεχνικής σκοπιάς να γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που έχουμε ήδη συμφωνήσει ε, και στα πλαίσια της Europol και στο σύστημα SIS, το σύστημα πληροφοριών Schengen, αλλά και σε άλλα συστήματα. Η ανταλλαγή αυτή θα πρέπει να γίνεται και σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι η ανταλλαγή για την οποία έχουμε συμφωνήσει μεταξύ των κρατών μελών της, Ένωσης, της Ένωσης δεν γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δεν ε, ε, ε, καταχωρούνται στο σύστημα οι πληροφορίες παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί και μετά δεν χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες στο σύστημα. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, διότι δεν έχει κανένα νόημα να αποθηκεύουμε απλώ στοιχεία ε, και να μην χρησιμοποιούνται μετά με τον κατάλληλο τρόπο. Πέραν αυτού, οι προτάσεις για την ενίσχυση της ε, νομικής δυνατότητας να συνδέονται τα συστήματα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους Κατά την άποψή μου θα πρέπει να περιορίζεται απλώ την ενίσχυση της δυνατότητας ελέγχου διαφορετικών συστημάτων ταυτόχρονα, εάν ε, Κάποιο μπορεί να ελέγχει διαδοχικά τα συστήματα, δηλαδή για να εξοικονομήσουμε κάποιο χρόνο. Εδώ όλοι θα πρέπει να συμφωνούν ότι θα πρέπει να γίνονται τέτοιε αλλαγέ. Αλλά η ενίσχυση τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτή κάθε αυτή ε, δεν ξέρω αν είναι σωστή, σα εφιστώ την προσοχή και δεν ξέρω και αν ε, υπάρχει προστασία δεδομένων. Διότι εκεί αλλάζει ο στόχος αυτών των συστημάτων και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με κάτι τέτοιο και να δούμε αν μπορούμε να ενισχύσουμε την δυνατότητα να εφαρμόζεται καλύτερα αυτό το οποίο είναι ήδη ε, νομικώς ε, εφικτό και ε, να, που έχουμε ήδη συμφωνήσει να κάνουμε. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σε συνέχεια των όσων ακούστηκαν είναι ότι υπήρξαν πολλές αποφάσεις του δικαστηρίου και προσφάτως και μία γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το τι είναι αναλογικό προκειμένου να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς ασφαλείας. Και πρέπει να πω ότι η γραμμή που έχει τηρήσει το δικαστήριο σε όλες αυτές τις αποφάσεις, ξεκινώντας από την απόφαση διατήρησης δεδομένων του 2014 και την γνωμοδότηση για την συμφωνία με το Καναδά για την ανταλλαγή του PNR τον Ιούλιο, είναι σαφής, απόλυτα σαφής. Και λέει ότι η αποθήκευση και συλλογή προσωπικών δεδομένων όλων των πολιτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να αιτιολογείται ε, άνευ λόγου, θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, να περιορίζεται χρονικά και να αφορά κάποιες συγκεκριμένες υποψίες ή κινδύνους ή κάποια ε, εγκληματική δραστηριότητα. Με Ό,τι κάνουμε λοιπόν για τη διαλειτουργικότητα θα πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε και τα συστήματά μας. Ιδάλλως, απλώς θα έχουμε συνεχώς συστήματα τα οποία ε, θα λειτουργούν παράνομα. Και κάτι ακόμα το οποίο προέκυψε από τη γνωμοδότηση για τα ε, PNR Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Τα εξοδετικά στοιχεία θα πρέπει να διαγράφονται όταν δεν χρειάζονται πλέον. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει ολοκληρώσει το ταξίδι του, για παράδειγμα. Και μόλις ε, ε, δημιουργήθηκε, όπως είπατε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα PNR και μόλις ε, ψηφίσαμε και το σύστημα εισόδου-εξόδου. Και σε κανένα από τα δύο συστήματα δεν υπάρχει ένδειξη ότι κάποιος μόλις ολοκληρώσει το ταξίδι του και δεν βρίσκεται σε κάποιο κατάλογο υπόπτων ή κινδύνου, θα πρέπει αμέσως να διαγράφονται τα στοιχεία του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί τώρα και θα ήθελα να ασχοληθείτε και με αυτό. Η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ πολύ. Μας υπενθυμίσετε κύριε Πρόεδρε ότι θέλουμε να έχουμε ευφυή σύνορα. Εγώ ε, δεν νιώθω άνετα με αυτή την ορολογία, δεν ξέρω τι είναι τα ευφυή σύνορα και δεν είμαι βέβαιη ότι η τεχνολογία κάνει τα πράγματα πιο ευφυή. Ε, μας λέτε κύριε Επίτροπε ότι ε, δεν είναι μεγάλος αδελφός όλα αυτά. Ακούω τι μας λέτε, αλλά πραγματικά αυτό που θα ήθελα να σας πω εξαρτάται από τον ε, καθένα, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι όλοι ισότιμοι ε, όσον αφορά αυτό το σύστημα. Έχουμε περίπου 15 κείμενα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλα οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ενίσχυση της ε, ασφάλειας, ναι, εγώ είμαι υπέρ της ενίσχυσης ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και δεν ξέρω ποιος το είπε, ότι το κείμενο είναι και τεχνικό και πολιτικό. Τουλάχιστον όμως ε, να μην ε, υπερτερεί το τεχνικό εις βάρος του πολιτικού στοιχείου και στα πολιτικά στοιχεία υπάρχει όλο και μεγαλύτερη σύγχυση και θα ήθελα να δείτε και την εξέλιξη της ορολογίας για αυτά τα ευφύ σύνορα από τότε που αρχίσαμε να τα συζητάμε αυτά τα ευφύ σύνορα. Είναι ένα αμάλγαμα όλο και περισσότερο ε, όρων που αφορούν την μετανάστευση και την τρομοκρατία. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η πλειοψηφία των δραστών των ε, τρομοκρατικών πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αλλοδαπή, αλλά ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Και επίσης θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα αυτής της ε, ε, προθύστερης στάσης με το ΕΤΙΑΣ. Το ΕΤΙΑΣ είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο θα αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση διαβατηρίου αλλά θα ζητάμε περισσότερες πληροφορίες από όσα ζητούμε τελικά από ανθρώπους που ε, λαμβάνουν θεώρηση διαβατηρίου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι τα δικαιώματα αυτών των υπηκών τρίτων χωρών δεν ε, προστατεύονται όταν τους ζητάμε ε, στοιχεία, για παράδειγμα, για την υγεία τους. Και θα ήθελα να ξέρω τι σχέση έχουν τα στοιχεία για την υγεία τους στο σύστημα αυτό. Και εδώ πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον για το ETIAS. Γιατί ε, εμπιστευόμαστε τη διαχείριση στο, ε, του ETIAS ε, στο Frontex και όχι στην Ιουλίζα. Διότι όπως είπατε και εσείς η Ιουλίζα είναι ο θεματοφύλακας της συνεκτικότητας των συστημάτων. Γιατί λοιπόν υπάρχει εξαίρεση, εξαίρεση και είναι η Frontex αρμόδια για το ETIAS. Ε, κάτι άλλο τώρα η εξάλληξη του SIS, του Συστήματος Πληροφοριών Schengen. Γιατί εξελίσσεται το σύστημα χωρίς πραγματική αξιολόγηση. Θα συμφωνήσω με κάποιον από τους προαλήσαντες που επέμενε αυτό σε αυτό το θέμα. Και γιατί έχουμε ένα εργαλείο για τις πολιτικές επιστροφέων και πάλι εις βάρον ε, των ενδιαφερομένων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες όντως έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Αντίθετα με τα όσα λέτε, συλλέγουμε ένα και περισσότερο στοιχεία και τα συλλέγουμε για, μία, ολοένα και, για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά και θα γίνονται όλο ένα και λιγότερο σεβαστά. Διότι στα κείμενα τα οποία μας υποβάλλεται δεν μπορούμε πλέον να καταλάβουμε και μέχρι ποιο βαθμό θα φτάνουν αυτές οι διατάξεις, διότι ε, τα κρύβεται όλα πίσω από τεχνικά επιχειρήματα. Πρέπει πραγματικά να αξιολογήσουμε την κατάσταση και έχουμε χρόνο κύριε Επίτροπε. Ακόμα και αν πρέπει να είναι σε λειτουργία τα συστήματα μέχρι το 2020, Τώρα είμαστε στο 2017. Έχουμε χρόνο να εκπονήσουμε και κάποιες μελέτες πριν ε, να είναι πολύ αργά. Και έχουμε και χρόνο να ε, θέσουμε τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους. Διότι καταλαβαίνω ότι ε, πρέπει ίσως να υπάρχει ανάγκη για τα θεσμικά όργανα και κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει προκειμένου να αμφισβητήσει τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη. Αλλά όσον αφορά τις συγκεκριμένε αρμοδιότητες, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα εφαρμόσουν. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς εφαρμόζουν ή μάλλον δεν εφαρμόζουν κάποιες διατάξεις και κυρίως ό,τι αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, δεν χρειάζεται τώρα να σας ε, αναφέρω παραδείγματα για τις χώρες οι οποίες ε, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, η Λαούρα Φεράρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Ε, θέλω να σας πω, είμαι ακράταντα πεπισμένη ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό το λέμε εδώ και καιρό. Και έτσι λοιπόν ε, με μεγάλη χαρά άκουσα την πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει αυτή η ενταλλαγή πληροφοριών. Ε, θα είμαι πολύ συγκεκριμένη στην ερώτησή μου. Δηλαδή, θα με ενδιέφερε να γνωρίζω πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το πώς θα λειτουργεί αυτή η διαλειτουργικότητα που αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών. Δηλαδή τελικά τι θα είναι, θα είναι ένα είδος υπερδομής, άλλη μία τράπεζα δεδομένων η οποία θα μαζεύει τα δεδομένα από τις τράπεζες που ήδη υπάρχουν ή μήπως θα είναι κάποιος ε, τεχνικός μηχανισμός ο οποίος θα συνδέσει μεταξύ τους ε, τις τράπεζες δεδομένων. Υπερδομή ή η ίδια σύνδεση των ήδη υπαρχούσων ε, τραπεζών δεδομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, και εμείς μελετήσαμε λιγάκι τη Συμφωνία του Δουβλίνου, τη Eurodac, ε, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι για να κατανοήσει κανείς κάποια πληροφορία είναι αγκασμένο να καταφύγει σε διάφορες τράπεζες δεδομένων. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή συντονισμός, ε, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει διασύνδεση των κείμενων ε, τραπεζών δεδομένων. Και όπως είπε και ο συνάδελφος κυρίως Άρμπρεχτ, δεν ε, υπήρξε ποτέ ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών άμεσα στα κρατημέλη για διάφορους λόγους, ε, γραφειοκρατικούς, διοικητικούς, αλλά μερικές φορές και δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, υπήρχε κάποια επιφυλακτικότητα. Εγώ λοιπόν θέλω να γνωρίζω το πώς είναι δυνατόν πρακτικά να λειτουργεί η διαλειτουργικότητα και ποιο είναι και το κόστος που θα συνεπάγεται η συντήρηση αυτής της πλατφόρμας ή αυτού του μηχανισμού αν θέλετε. Η Μπάρμπαρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αβραμόπουλε. Ε, πολύ ιδιαίτερα διεξοδικά τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας και κύριε Γκάρκοφ, ευχαριστούμε πολύ και για τις ε, δικές σας τις πληροφορίες. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια κατάσταση όπου η αρμόδιοι δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ε, λόγω του ότι υπάρχει τεχνικός περιορισμός. Έχω την εξής ερώτηση. Η έβδομη έβδομη έκδοση πρόοδου προς μια αποτελεσματική και ασφαλή ένωση αναφέρεται στο γεγονός ότι οι ομάδες εμπειρογνωμών, σχετική έκθεση δηλαδή δεν κατέδειξαν ότι είναι απαραίτητο να ελέγχονται όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέπτεται να εξετάσει την καταγραφή ανθρώπων ε, που ζουν, ε, που ταξιδεύουν έτσι ώστε να εντοπιστούν ε, κάποιοι ύποπτοι οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε τρομοκρατικές ενέργειες. Όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα και σε σχέση με την ασφάλεια, η Κομισιόν έχει επιτυχεί κάποια πρόοδο. Και όσον αφορά στη διαλειτουργικότητα, έχω μία ερώτηση την εξής. Πότε ακριβώς πιστεύετε ότι θα επιτύχουμε τη διαλειτουργικότητα από διοικητικής ε, και διαχειριστικής πλευράς, τεχνικής περισσότερο πλευράς. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Φερέρα, ποια είναι η χώρα εκείνη η οποία ενδεχομένω δεν επιθυμεί να συνεργαστεί και γιατί. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά. Η Μαρή Λάουριστεν. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημά μου στρέφεται προς τον κύριο Γκάρκοφ. Υποθέτω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να ακούσουμε τις ε, γενικές ε, δηλώσεις, τις ε, πολιτικές δηλώσεις. Η Γιουλίσα είναι πραγματικά ένα τεχνικό εργαστήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εφαρμογή όλων αυτών των γενικών αρχών που προετοιμάζουμε εδώ από κοινού. Θα ήθελα λοιπόν ε, να θέσω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, σε σχέση με την ασφάλεια και άλλα θέματα και αυτό που με ενδιαφέρει κύριε Γκάρκοφ είπατε ότι η διαλειτουργικότητα είπατε ότι η προστασία των δεδομένων καθίσταται καλύτερη μέσω της διαλειτουργικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντική δήλωση, είναι πολύ σημαντικό αν μπορείτε να μας το αποδείξετε κιόλα, ε, να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα πώς γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξή. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε κάποιους κανόνες ε, στο πλαίσιο της νομοθεσίας μας και επιζητούν ανάλυση κινδύνου. Έχει γίνει κάτι τέτοιο, μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιοι ήταν οι κυριότεροι κίνδυνοι τους οποίους εντοπίσατε στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής της εφαρμογής διαλειτουργικότητας. Και το δεύτερο ερώτημα όταν ε, εντοπίζετε τους κινδύνους, ε, είπατε ότι ήρθατε σε επαφή με τον επόπτη προστασίας δεδομένων και θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν τα βασικά σημεία επί των οποίων ε, διαβουλευθήκατε και πώς πήγε αυτή η συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βίνπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Αβραμόπουλο τα ισχυρότερα και ευφιέστερα συστήματα πληροφορικής ε, πράγματι είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Σε αυτό συμφωνώ απολύτω. Συμφωνώ με πολλούς ε, όσους πήραν το λόγο και είπαν ότι χρειάζεται καλύτερο συγχρονισμός μεταξύ ε, των συστημάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επεξεργαστούμε. Και αυτό το θέμα του Big Brother, του μεγάλου αριθμού που σε παρακολουθεί, νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει κάποιο είδους παρακολούθηση, κάποιο είδους ε, επίβλεψη. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να ε, με, ε, να με πάρει κανείς ε, στην κάμερα όταν ε, παίρνω λεφτά από ένα ATM για παράδειγμα. Κάποιοι όμως έχουν πρόβλημα με αυτό. Το PNR είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα και το υπερψηφίσαμε. Το θέμα είναι πότε θα λειτουργήσει. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συχνά αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι με κακές ε, προθέσεις ε, περνούν στις χώρες μας, ε, ο κόσμος μπαίνει σε πολύ μεγάλους αριθμούς πλέον στις χώρες μας και αυτό που ίσως θα έπρεπε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τα δικά μας τα, σύνορα. Τι νόημα έχει να έχουμε συστήματα αν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτού του ανθρώπους που σε τεράστιου αριθμούς ε, περνούν τα σύνορά μας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς το σύστημα θα αντιμετωπίσει το θέμα, ας πούμε, των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στο αεροπλάνο δεν είναι και ανόητη στο κάτω-κάτω τη γραφή. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι στα σύνορα, γιατί για την ώρα δεν λειτουργούν καλά. Και αναφέρεται από τον Νοέμβριο δεν θα γίνονται πια έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κινίτσι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Επίτροπο Αβλαμόπουλο και τον Διευθυντή τον κύριο Γκάρκοφ για την παρουσία τους και την εισαγωγή που έκαναν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για την ασφάλεια των χωρών μας. Προσωπικά σας το είπα επανειλημμένος, εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη συνεργασία και επομένω την ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς ασφαλείας. Και ε, προφανώς και είμαι ε, καθόλου ε, υπέρ της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών. Θα ήθελα όμως να παρουσιάσω κάποιες πρώτες σκέψεις ε, και μία ερώτηση γενικού χαρακτήρα από εκεί και πέρα. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε σε ε, περιβάλλον εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών, το οποίο οικοδομείται τον τελευταίο καιρό ε, και ίσως και λόγω των τρομικρών, τρομοκρατικών επιθέσεων που δυστυχώς έπληξαν κάποιες χώρες και επομένως κατέδειξαν όλο και περισσότερο την ανάγκη ασφάλειας και συνεργασίας στον τομέα αυτό και διαπιστώσαμε δυστυχώς και κάποιες ελλείψεις, ε, ιδίως ε, λόγω κάποιων τρομοκρατικών επιθέσεων ε, στην ανταλλαγή πληροφοριών. Εκτιμώ λοιπόν την ιδέα της διαλειτουργικότητας η οποία θα αποτελέσει και μία ενιαία δικτυακή πύλη, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι, ε, να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση για όλες τις δυνάμεις της αστυνομίας, τις δυνάμεις της τάξης, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ασφαλείς οι χώρες μας. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Εάν θεωρήσουμε ότι όντως η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να έχουμε καλύτερη χρήση από πλευρά κρατών μελών των βάσεων δεδομένων. Ακριβώς ε, λόγω αυτού του προφίλ της ε, δημιουργίας ενός ε, περιβάλλοντος εμπιστοσύνης. Θα μπορέσει να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, τις επικρίσεις που είχαμε και που ορισμένες φορές δεν επέτρεψαν και στην την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Τι μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατάσταση κατεύθυνση, ε, να παρέχουμε πόρους, εκπαίδευση, κατάρτιση, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Και τώρα προς τον Διευθυντή τον κύριο Γκάρκοφ ε, δύο σκέψεις και μία ερώτηση τρόπον τινά. Ε, πολύ σωστά αναφερθήκατε στην ανάγκη και μέσω του συστήματος της διαλειτουργικότητας των ε, πληροφοριών να έχουμε εσωτερική ασφάλεια, διαχείριση των συνόρων, διαχείριση της μετανάστευσης και το καθεξής. Ε, στο θέμα αυτό λοιπόν, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν και εγγυήσεις και σεβασμός των πολιτών όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα για την ιδιωτική του ζωή. Στο θέμα της μετανάστευσης θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες περαιτέρω σκέψεις ε, για τα αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να έχουμε μέσω της χρήσης ενός συστήματος διαλειτουργικότητας των δεδομένων. Και τέλος, αυτή είναι μια ερώτηση ίσως πιο συγκεκριμένη, εάν η πόρη του Ιγιουλίσα, ε, εγώ θα είμαι και σκιώδης εισηγήτρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για το νέο σας κανονισμό, η πόρη σα, όχι τόσο οικονομική αλλά γενικότερα οι πόροι σα ε, που απαιτούνται για να έχετε ένα αποτελεσματικό σύστημα, επαρκούν ή ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να επενεξετάσουμε κάποια σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ιάννα Γκόμες. Ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τον κύριο Γκάρκοφ για την παρουσία τους εδώ σήμερα και για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Οι ερωτήσεις μου αφορούν τη λειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα, κυρίως τη λειτουργικότητα του ίδιου e Όταν ε, Ε, καταλαβαίνω όλα αυτά που είπατε για την ε, προστασία των δεδομένων, να είναι περιορισμένο ο σκοπό του, να υπάρχει διαλειτουργικότητα του συστήματο, αλλά δεν θα είναι ο μεγάλο αδελφό. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται όμως όταν η φραγμή στη διαλειτουργικότητα δεν είναι τεχνικής φύσεως, αλλά είναι πολιτικής φύσεως. Έστω, για παράδειγμα, η πιο πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελόνη. Εκεί επισημάναμε ότι η αστυνομία της ε, Βαρκελόνης, ε, της Καταλωνίας, δεν είχε πρόσβαση στις πληροφορίες για τους τρομοκράτες ε, που, που οργάνωσαν και εξετέλεσαν την επίθεση. Πληροφορίες οι οποίες διατίθεταν από τα άλλα κράτη-μέλη και ήταν διαθέσιμα μέσω Ευρωπόλ. Επομένως, το πρόβλημα και πάλι, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολιτική φραγμή εντός των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών, ε, για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Το ίδιο ισχύει και με το PNR. Λυπάμαι κύριε Επίτροπε, αλλά τα κράτη-μέλη βιάστηκαν να κατηγορήσουν το Κοινοβούλιο γιατί δεν ενέκρινε το PNR και τώρα τα κράτη-μέλη καθυστερούν την εφαρμογή του συστήματο ανταλλαγή στοιχείων επιβατών. Και ξέρουμε ότι το PNR έχει πάρα πολύ σημαντικά κενά εάν θέλει να πετύχει το σκοπό για τον οποίο ψηφίστηκε. Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνονται οι πτήσει τσάρτερ γιατί δεν τις ήθελαν τα κράτη-μέλη, όχι γιατί το Κοινοβούλιο δεν τι πρότεινε και γιατί για παράδειγμα, για τα ιδιωτικά αεροπλάνα. Οποιοςδήποτε Σαουδάραβας πρίγκιπας ή μη μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα και να πάει στις ακτές μας ή σε άλλες ενδιαφέρουσες τοποθεσίες και ταξιδεύουν με το ε, αεροπλάνο τους όπου θέλουν. Ε, και μπορεί να μεταφέρουν και φορτίο ή χρήματα. Ποιο ελέγχει, κανεί δεν ελέγχει και κανένα δεν υποτίθεται ότι θα τα ελέγχει αυτά όλα. Και μετά, έχω και την εξή ερώτηση. Υποθέτουμε ότι οι τρομοκράτε έρχονται από το εξωτερικό, αλλά αυτοί οι οποίοι μα επιτίθηκαν είναι δικοί μα πολίτε. είναι εκ των έσω. Πού είναι λοιπόν η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και πού επενδύεται σε προγράμματα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και τη, ε, τον εντοπισμό των ε, ε, ριζοσπαστικοποιημένων που σημαίνει ότι πρέπει να βοηθήσουμε και τις κοινότητες από τις οποίες ε, προέρχονται αυτοί οι τρομοκράτες. Τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να σταματήσουμε να εισάγουμε οι μάμιδες που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καθοδηγητές ε, και οργανώνουν ε, τρομοκρατικές επιθέσεις. Και κάτι τελευταίο. Εγώ συμμετείχα σε αυτή την ομάδα Σέγγεν, στην οποία επικεφαλής ήταν ο συνάδελφος ο Κάρλος Κοέλιο και ε, τι κάνουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις που διαπιστώσαμε και δεν πρόκειται σίγουρα για ένα κράτος μέλος ότι θεωρήσεις διαβατηρίων ε, οι οποίες κανονικά δεν έπρεπε να είχαν δοθεί τελικά δόθηκαν, κανείς δεν κατανοεί γιατί και η ε, ε, εξήγηση είναι ότι πρόκειται περί διαφθοράς του συστήματος και ε, αφορά και τα σύνορα την απόφαση να εκχωρηθεί μια θεώρηση διαβατηρίων. Όταν τα κράτη-μέλη λοιπόν προωθούν τη διαφθορά μέσω ενός σύστηματος ε, επενδύσεων και χρυσές θεωρήσεις διαβατηρίων, μπορεί κανείς να κατηγορήσει μικρά γραφεία που δίνουν απλώς ε, θεώρηση διαβατηρίου Σέγγεν όταν κανονικά δεν θα επιτρεπόταν να τους δοθεί και ξέρετε σε ποια χώρα να φέρουμε. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντ, ε, και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Ευχαριστώ τον Διευθυντή κύριο Γκάρκοφ. Εγώ θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί είδα ότι αυτό, αυτό το καλοκαίρι επισκέφτηκα το hot spot στον Τάραντο και μίλησα διαμακρών και με τη Europol σχετικά με την ε, διατήρηση και διαφύλαξη των δεδομένων. Είδα λοιπόν ότι στο Τάραντο ε, τα δεδομένα συγκεντρώνονται και ανταλλάσσονται και με άλλους φορείς. Η δική μου ερώτηση αφορά τη διαλειτουργικότητα. Ε, δηλαδή αυτή η διαλειτουργικότητα πώς θα λάβει η χώρα. Ε, θα υπάρχει σεβασμός των δεδομένων, θα υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, για να κατανοήσω κατά πόσον θα αποφευκτεί αυτή η σχέση ανάμεσα στη μετανάστευση και την τρομοκρατία, είναι ε, μια ορολογία που χρησιμοποιείται σχεδόν ευρέως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ λοιπόν αυτό που βιώνουμε είναι πόλεμος είναι πραγματικός πόλεμος και κάποιος ε, πρέπει να τον αναχαιτήσει. Μερικές φορές τον πόλεμο μπορεί κανείς να τον αντιμετωπίσει με εκπαιδευτικά εργαλεία. Έχουμε την, ε, το κυνήγι του ξένου, αυτό που ζούμε σήμερα. Κανείς δεν γράφει πάνω στο κορμί του ότι ήρθε χτες ή σήμερα. Μπορεί να έχει έρθει και πριν από 20 ολόκληρα χρόνια. Και αυτή λοιπόν η σύγκρουση νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επιτέλους αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε που ήσασταν ε, σύντομη Σεσίλια. Και τέλος, ο κύριος Λοπέζ Αγγιλάρ. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονός ότι είμαι και ο τελευταίος που λαμβάνει το λόγο, ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα βεβαίως κύριε Επίτροπε και κύριε Γκάρκοφ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, που ε, μας μιλήσατε για τη σημασία της διαλειτουργικότητας. Θέλω όμως επίσης να πω ότι κατά την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι όσοι πήραν το λόγο είπαν το σωστό, ότι όλοι ανησυχούμε. Ανησυχούμε για τη σημασία που έχει το ε, να ε, μπορεί κανείς ε, να διασφαλίσει την ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Και θα ήθελα να κάνω και δύο άλλες ερωτήσεις, δύο πραγματικές ερωτήσεις. Πρώτον, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να υπάρχει πραγματική ε, διαλειτουργικότητα ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί αυτό έλειπε τα τελευταία χρόνια. Κατά τα άλλα, ποιες είναι οι ελλείψεις, οι αντιστάσεις, ε, τα εμπόδια που ε, παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη και για ποιους λόγους, γιατί δεν είναι το ίδιο να αντιμετωπίζει κανείς ε, θέματα ασφάλειας από θέματα εθνικής ασφάλειας, ατομικής από εθνική ασφάλεια. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει λόγω του ότι ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το οποίο δικαστήριο επισημαίνει ότι κάθε φορά που προσπαθούμε να επιβάλλουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαχείριση των πληροφοριών κάθε φορά ξεπεράσαμε τα όρια του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όπως ακριβώς φάνηκε και με την τελευταία απόφαση για το Καναδικό Ευρωπαϊκό ε, PNR. Πρόεδρος και Επίτροπε. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις ε, και νομίζω ότι παρουσίασαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις ε, παρεμβάσεις σας, ε, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας, αλλά και τις σκέψεις σας. Πράγματι, όλες δείχνουν ότι συμφωνούμε ως προς την αρχή, την αρχή την οποία μόλις τόνισε ο κύριος Λόπες Αλγκυλάρ, Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας. Αυτό είναι το κύριο καθήκον μας, χωρίς βέβαια να υπονομεύουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικότερα το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων. Ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε ένα νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων το οποίο θα αρχίσει να ισχύει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αρχές που συμπεριλαμβάνει είναι οι κατευθυντήριες γραμμές μας, είναι οι ο γνώμονάς μας ως προς την εφαρμογή της ε, διαλειτουργικότητας. Ε, Μέτσολα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ε, για την υποστήριξή σας έχετε απόλυτο δίκιο. Τα συστήματά μας πρέπει να συνδέονται καλύτερα, αλλά πρέπει και να χρησιμοποιούνται καλύτερα. Αυτό είναι ακόμη σημαντικό, όπως είπε και η κυρία Ζήπελ. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της ε, διαλειτουργικότητας είμαστε υπέρ της ε, προσέγγισης της, του clean desk approach, δηλαδή θέλουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα εργαλεία ε, τα οποία ε, έχουμε ε, στη διάθεσή μας, όπως το σύστημα εισόδου-εξόδου και το σύστημα πληροφοριών της Engen, το SIS. Πράγματι, το να κάνουμε μία αξιολόγηση όλων αυτών των συστημάτων πριν ε, αρχίσει η διαλειτουργικότητα θα ήταν πολύ δυσκολότερο. Αυτή τη στιγμή ε, θα αρχίσουν να ισχύουν τα συστήματα αυτά, θα αρχίσει και η διαλειτουργικότητα. Θα κάνουμε μία ε, λεπτομερή μελέτη επιπτώσεων για την πρόταση διαλειτουργικότητας και βέβαια θα λάβουμε υπόψη και τις πτυχές προστασίας των δεδομένων. Όσον αφορά τώρα την πρόοδο της ομάδας ε, εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπόδου, ο ε, διευθυντής της Ιουλίσα θα σας πει περισσότερα. Κυρία Ζίπελ και κυρία Όλμπριχτ. Όσον αφορά το, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά ως προς το PNR, καταρχάς, η απόφαση του Ευρωπαϊκού του Δικαστηρίου ε, ε, ε, αναφέρει ότι το PNR πρέπει να θέτει τις νομικές παραμέτρους οποιασδήποτε μελλοντική συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών. Είναι πραγματικά ένας πολύτιμος οδηγός για το πώς θα προχωρήσουμε. Η απάντηση του Δικαστηρίου κατόπιν δικού σας αιτήματος είναι η προτινόμενη συμφωνία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα μορφή της, γιατί κάποιες από τις διατάξεις της είναι μη συμβατές με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ειδικότερα το δικαίωμα ε, για την προστασία δεδομένων ε, και ε, τον ιδιωτικό βίο. Το δικαστήριο αναγνώρισε πράγματι ότι η μεταφορά δεδομένων PNR από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Καναδά δικαιολογείται ο, μόνο για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, ή την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών. Όμως, κάποιες διατάξεις της προτινόμενης συμφωνίας δεν ε, περιορίζονται σε αυτό που αυστηρά είναι απαραίτητο και δεν ε, αναφέρουν ρητά συγκεκριμένους κανόνες. Δεδομένου λοιπόν ότι η χρήση των δεδομένων PNR είναι σημαντική για να καταπολεμήσουμε το σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία, εμείς θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συνεχίσουμε τη μεταφορά των δεδομένων PNR, ψευόμενοι πλήρως ε, την απόφαση του ε, δικαστηρίου ε, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εμείς ολοκληρώνουμε την ανάλυση μας ως προς την νομοδότηση του δικαστηρίου. Θα ζητήσουμε και σχετική εντολή σύντομα από το Συμβούλιο για να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες με τον Καναδά για μια βελτιωμένη συμφωνία η οποία θα συνάδει πλήρως με τις απαιτήσει που αναφέρονται στην γνωμοδότηση του δικαστηρίου. Όσον αφορά τώρα τις συνέπειες για τη διαλειτουργικότητα, η άποψη του δικαστηρίου δεν εφαρμόζεται πλήρως ε, για τη διαλειτουργικότητα των ε, συστημάτων ε, πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συστημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όμως θα αναλύσουμε τις ευρύτερες συνέπειες της διαλειτουργικότητας για μεγάλης κλίμακα συλλογή δεδομένων και βεβαίως αυτό θα αφορά και τη διαλειτουργικότητα οι δικές μας επιλογές πολιτικής για τη διαλειτουργικότητα θα σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και βεβαίως και την προστασία δεδομένων. Θα εξασφαλίσουμε ότι κάθε πρόταση που θα γίνει θα συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις ε, που έχει θέσει ε, στην ε, στις αποφάσεις του αλλά και στη γνωμοδότησή του το δικαστήριο ως προς το PNR προσφάτως. Συμφωνώ απολύτως ε, κύριε Όλμπριχτ με το θέμα που θέσατε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει διασύνδεση των συστημάτων. Πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι η επιλογή που είναι πιο φιλική προς την προστασία των δεδομένων. Κυρία Ζήπελ, εγώ καταλαβαίνω, ε, γνωρίζω ε, το αίτημά σας για ε, την πρόσβαση στα δεδομένα. Οι υπηρεσίες μου έχουν βασιστεί στον κανονισμό 49 του 2001 ε, σε μοικές περιπτώσεις ε, τμήματα της αλληλογραφίας ε, έχουν διαγραφεί βάσει νόμου. Η πρόσβαση δεν έγινε δεκτή λόγω ε, προστασίας ε, της ε, διαδικασίας εσωτερικής, εσωτερικής διαδικασίας αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο διαμεσολαβητής βεβαίως θα μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να διαλευκάνουμε αυτό το ζήτημα. Τα μελλοντικά μας συστήματα θα ε, είναι προσπελάσιμα, ε, θα συμπεριλαμβάνουν πηγές όπως βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα ταυτότητας και θα είναι διαλειτουργικά. Όμως αυτό δεν θα γίνει εις βάρος της προστασίας δεδομένων. Αντιθέτως, όλες οι δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των ε, δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων, θα συμπεριληφθούν στις μελλοντικές μας προστάσεις. Ο έλεγχος της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, στα δεδομένα αυτά βεβαίως έχουν ε, μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη σημασία και θα γίνει βέβαια σύμφωνα με τους κανόνες περί δεδομένων και θα ε, περιορίζεται στο σκοπό που εξυπηρετεί κάθε σύστημα. Ο έλεγχος της πρόσβασης μπορεί και θα επιθευθεί μέσω ε, του σχεδιασμού του λογισμικού για το κάθε σύστημα. Καταρχάς, ε, θα συνεργαστούμε με τις αρχές προστασίας δεδομένων κατά την προετοιμασία των ε, μελλοντικών μας πρωτοβουλειών. Τα ε, συστήματα τεχνολογίας και τα συστήματα πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων της ασφάλειας και της μετανάστευσης μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα ε, μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων ε, και μέτρα ε, αποκατάστασης θα είναι τμήμα των προτάσεών μας στο μέλλον και η πρότασή μας περί διαλειτουργικότητας θα το λάβει αυτό υπόψη πλήρως. Η, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ε, είναι, υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων ε, που θα συνάδει πλήρως ε, με τους επικαιροποιημένου κανόνες προστασίας δεδομένων και θα υπάρχει βέβαια μία πολύ περιορισμένη, αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα. Κυρία Βερζιά, είπατε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχει να κάνει με την καταπολέμηση της ρίζος παστικοποίησης ε, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, διαφορετικό αλλά πολύ σημαντικό και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε σύντομα και με την κυρία Γκόμες ε, όσον αφορά το ΕΤΙΑΣ. Όσον αφορά το ετιάς δεν ζητάμε περισσότερες πληροφορίες ε, ε, ως προς αυτό ε, από ό,τι για τις θεωρήσεις. Ε, συλλέγουμε πολύ λιγότερα δεδομένα. Για παράδειγμα, δεν συλλέγουμε βιομετρικά δεδομένα όσον αφορά την έγκριση και την εφαρμογή είμαι πεπισμένος ότι ε, δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας γιατί μας ξεπερνούν οι εξελίξεις και μερικές εξελίξεις είναι πραγματικά δραματικές, ε, λαμβάνουν χώρα πολύ πιο γρήγορα από τις δικές μας αποφάσεις, δεν μπορούμε να τις προλάβουμε και δεν μπορούμε να, να, να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η εφαρμογή και η καλή χρήση του συστήματός μας είναι κρίσιμη σημασία και είναι κάτι που το είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια. Για σας, κυρία Φεράρα, η διαλειτουργικότητα. Θα κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή τα συστήματά μας θα μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει για αναζήτηση, να υπάρχει μόνο μια δικτυακή πόλη αναζήτησης. Δηλαδή μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από όλα τα υπόλοιπα μεμονωμένα συστήματα και βιομετρικές πληροφορίες αλλά και αλφαριθμητικά στοιχεία δεν ε, δημιουργούμε μία ε, βάση δεδομένων πολύ μεγαλύτερη που να τις συμπεριλαμβάνει όλες. Η καταγραφή όλων όσων ε, διέρχονται τα σύνορά μας θα έχει σημαντικές συνέπειες ως προς την προστασία δεδομένων και γι' αυτό το λόγο η έκθεσή μας ε, για την ε, ε, Ένωση της για την ασφάλεια της Ένωσης μας έδειξε ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά. Κυρία Κινίτσι, τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν μυστικές πληροφορίες, ε, ενδεχομένω εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια κράτη-μέλη ε, συνεργάζονται ε, όντω ανταλλάσσουν πληροφορίε. Εμεί όμω θα θέλαμε όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Η αρμοδιότητα τη Ένωση αναφέρεται ρητά ω προ αυτό στι συνθήκε. Η εθνική ασφάλεια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Και όντως πρέπει να σημειώσουμε περισσότερη πρόοδος προς αυτό στο μέλλον τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι διαθέσιμα ε, στις ε, υπηρεσίες ασφαλείας και στις μυστικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ασφαλείας μπορούν επίσης να κάνουν καταχωρήσεις στο ΣΥΣ όσον αφορά υπόπτους τρομοκρατίας και κάποιες υπηρεσίες ασφαλείας όντως συνεργάζονται με την Ευρωπόλιδη. Και μάλιστα καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, γιατί αυτή τη στιγμή, δύο χρόνια μετά τα πρώτα δραματικά γεγονότα, δεν είμαστε πια στο ίδιο σημείο που ήμασταν τότε. Ε, εγώ δεν είχα τότε την ίδια εντύπωση και την ίδια αίσθηση που έχω τώρα σε σχέση με τη συνεργασία με την Ευρωπόλ. Όμω αυτή η συνεργασία με την Ευρωπόλ πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, ε, αυτή είναι η άποψή μου και τη μοιράζομαι μαζί σας μήπως έχει φτάσει επιτέλου η χρονική στιγμή να είμαστε τολμηροί και φιλόδοξοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ταμπού περί ασφάλειας του παρελθόντο και να συνεργαστούμε για να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα μυστικών πληροφοριών. Εγώ νομίζω ότι κάποια κράτη-μέλη δεν θα συμφωνήσουν με την ιδέα αυτή. Πριν από δύο χρόνια, όταν το είπα αυτό στην ε, δήλωσή μου, άκουσα τις πρώτες ε, αντιδράσεις, δύο χρόνια ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες ε, που είναι σε θέση να το συζητήσουν. Ίσως έχει περάσει ο καιρός και έχουν οριμάσει οι απόψεις. Ίσως αν υπήρχαν κάποιο, κάποιες τέτοιες πληροφορίες, αν υπήρχε μια τέτοια υπηρεσία ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να είχαμε προλάβει κάποια από αυτά τα δραματικά γεγονότα. Όμω αυτό είναι μια πολιτική δήλωση και νομίζω ότι το ε, βαθύ κράτος αντιστέκεται ε, σε αυτό. Πάντως, εδώ μιλούμε ούτω ή άλλω για την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποια μπορεί να είναι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το να μην υπάρχουν διακρίσεις. Όλοι οι πολίτες μας ε, και ειδικότερα όσοι βρίσκονται στα εξωτερικά μας σύνορα πρέπει να δείχνουν σεβασμό σε κάθε άτομο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ως μήνυμα θέλουμε να το στείλουμε παντού και δεν πρόκειται να σταματήσω να το επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε και δεν θα έπρεπε να μπερδεύουμε τους ε, μετανάστες με τους τρομοκράτες. Το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί πρέπει να εξουδετερώσουμε αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο ε, αυτή την τον επικίνδυνο λόγο. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την κοινωνία μας ότι, και μιλώ κυρίως για τους υπηκόους τρίτων χωρών ε, που ζουν μαζί μας, έχουν έρθει στις χώρες μας και δεν συμφωνούν καθόλου με τις ιδέες και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που διέπραξαν αυτά τα φρικτά εγκλήματα. Όπως είπα, το χρονοδιάγραμμά μας, ε, κύριε Αγγιλάρ, για, το, για την διαλειτουργικότητα είναι να κατατηθεί μια πρόταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο στόχος μας θα είναι να εγκριθεί και να εφαρμοστεί μέχρι το 2020. Και πράγματι οι αποφάσεις ε, του δικαστηρίου για ε, την ε, επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων θα αποτελέσει το γνώμονά μας καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Δημήτρη. Ο κύριος Γκάρκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Επίτροπος, καταρχάς ξεκινώντας από τις ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Ζίπελ για την αύξηση των βάσεων δεδομένων χωρίς να βελτισιοποιήσουμε απαραίτητο ε, τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. Στην πραγματικότητα κάνουμε και τα δύο. Η αύξηση των νέων βάσεων δεδομένων που προτείνεται στόχο έχουν να συμπληρώσουν ε, υφιστάμενα κενά πληροφοριών, κυρίως στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ σημαντική δουλειά για να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των υφιστάμενων ε, βάσεων δεδομένων. Παραδείγματο χάρη, το 2016 το ΣΥΣ χρησιμοποιήθηκε πάνω από 4 δις φορές σε σχέση με δύο ε, χρόνια πριν που η χρήση ήταν πολύ λιγότερη το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία τα οποία ε, καταχωρήθηκαν στο σύστημα. Το αυτό ισχύει και για άλλα συστήματα. Έγιναν προσπάθειες για να βελτιωθεί και η ποιότητα των δεδομένων ε, στα συστήματα, τα οποία συνεισφέρει ιδιαίτερα στην προστασία δεδομένων και στην ιδιωτικότητα. Για την ε, ποιότητα των δεδομένων ε, ένα λάθος θα μπορούσε να οδηγήσει και σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γι' αυτό και ε, έγινε η βελτίωση. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε τη διαλειτουργικότητα και εσείς νομίζετε ότι είναι διασύνδεση. Δεν είναι διασύνδεση. Η διασύνδεση σημαίνει ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ βάσεων δεδομένων. Διαλειτουργικότητα σημαίνει να μπορεί κάποιος να διαβουλευτεί διάφορες βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα. Ο στόχος είναι σαφής δεν θέλουμε και δεν θα εφαρμόσουμε τη διαλειτουργικότητα ε, εάν υπάρχει ανάγκη, θα αναλύεται ένα περίπτωση. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωσιοποιήσουμε και να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις βάσεις δεδομένων μέσω διαλειτουργικότητας, δηλαδή κάποιος να μπορεί να συμβουλεύεται τις βάσεις δεδομένων. Υπήρχε και μία ερώτηση για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαλειτουργικότητα. Με δύο λόγια, θα συνδέει τις βάσεις δεδομένων και θα επιτρέπει να ε, γίνεται ε, εξέταση των βάσεων δεδομένων με πιο απλό τρόπο, φυσικά ε, και βάσει του σκοπού για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί και τα δικαιώματα πρόσβασης τα οποία παρέχονται ε, συγκεκριμένα σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαλειτουργικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σαφής εδώ. Εδώ συνεργαζόμαστε προκειμένου η πρόταση για την ε, ο κανονισμό για τη διαλειτουργικότητα να υλοποιηθεί εντός του έτους και ελπίζουμε ότι θα μας δώσει και το χρονοδιάγραμμα που ο στόχος του είναι κατά βάση το 2020. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σας αναφέρω ότι οι προτάσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ε, για το ΕΤΙΑΣ ε, έχουν πολύ σημαντικά στοιχεία διαλειτουργικότητας ήδη ενσωματωμένα. Ε, θα είναι μια μακρά διαδικασία λοιπόν, ένα μακρύ ταξίδι το οποίο θα διαρκέσει πολύ αλλά αξίζει τον κόπο διότι τα αποτελέσματα θα είναι επωφελή για την εσωτερική ασφάλεια και για καλύτερη διαχείριση των συνόρων. Τώρα, για την ερώτηση της κυρίας Λόριτσεν και πώς θα ενισχύσουμε ε, τα συστήματα μέσω της διαλειτουργικότητας, χωρίς να επισέλθω σε πολλές τεχνικές ε, ε, λεπτομέρειες. Καταρχάς, έχουμε δύο πράγματα. Καλύτερη διαχείριση ταυτότητας, διότι αυτή τη στιγμή τα συστήματα τα έχουμε δημιουργήσει και τα διαχειριζόμαστε σε σιλό και αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα με διπλές ταυτότητας. Παραδείγματος χάρη, η τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο πέρσι τα Χριστούγεννα, οι υπηρεσίες εκεί διαπίστωσαν ότι ο επιτιθέμενος είχε 14 διαφορετικές ταυτότητες σε διαφορετικά συστήματα. Με τη διαλειτουργικότητα δεν θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και επίσης βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, διότι όπως αναφέρθηκε, όσο καλύτερη ποιότητα έχουν τα δεδομένα, τόσο πιο πιθανό είναι να υπάρχει παραβίαση ε, ατομικών δικαιωμάτων με τη χρήση των δεδομένων. Η ανάλυση κινδύνου της διαλειτουργικότητας είναι ευρύ θέμα και συνήθως η ανάλυση κινδύνου γίνεται σε ευρύ πλαίσιο. Θα ήθελα εδώ να σας καθησυχάσω. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία αφορά τη διαλειτουργικότητα ή περιλαμβάνει τη διαλειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου ή του αίτιας ε, ή το ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή εξοδου η Πύλη Αναζήτησης, υπάρχει ανάλυση κινδύνου και ε, βασίζεται σε συγκεκριμένα ε, και βάσει με την ανάλυση κινδύνου υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Άρα γίνεται αυτό ε, συστηματικά από τον Ιουλίσα. Ο Ιουλίσα επίσης συνεργάζεται στε, ε, στενά με τον Ευρωπαίο Πόπτη Προστασία Δεδομένων. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε τη συνήθι συζήτηση για τη διαλειτουργικότητα και κάποιε πτυχέ που αφορούν ε, ένα αποθετήριο κεντρικών δεδομένων, ε, όπω επίση ε, οργανισμού και υπηρεσίε που τακτικά ε, ελέγχονται από τον επόπτη δεδομένων. Επομένως αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι ε, τακτική και λαμβάνουμε υπόψη και τις συστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τις εκθέσεις εφαρμογής ε, στα διάφορα συστήματα. Επίσης, ο επόπτης προστασίας δεδομένων συμμετέχει και στην εξέταση του ΕΤΙΑΣ για την εφαρμογή των αρχών από το σχεδιασμό του συστήματος ήδη. επομένω, η προστασία των δεδομένων λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Η κυρία Κινίτσι ε, αναφέρθηκε στη σημασία να εγγυηθούμε προστασία δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητα. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η διαλειτουργικότητα δεν θέλει να αλλάξει τους κείμενους κανόνες πρόσβασης των δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα συμβουλεύεται κανείς τις βάσεις δεδομένων. Επομένως, η ιδιωτικότητα και η προστασία δεδομένων θα γίνονται σεβαστές με τον ίδιο τρόπο όπως και σήμερα, αλλά επίσης ταυτόχρονα η διαλειτουργικότητα προσφέρει καλύτερη εργαλειοθήκη για να ενισχύσουμε την προστασία δεδομένων και τις δικλείδες ασφαλείας για την ιδιωτικότητα. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, η κυρία Χινίτση αναφέρθηκε στους πόρους που έχει στη διάθεσή τη το Ιουλίσα. Η ε, διαλειτουργικότητα είναι τεράστιο καθήκον, τεράστια επιχείρηση, επομένως σίγουρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας, ώστε να μπορέσουμε να ε, διεκπαιρεώσουμε και τα θέματα της διαλειτουργικότητας όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα τα οποία έχουμε στην αναθεωρημένη εντολή μας. Και πιστεύω ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό για τη διαλειτουργικότητα θα ληφθούν αυτά υπόψη και θα ενισχυθεί ο οργανισμός ώστε να μπορέσουμε να ε, δώσουμε γέρος μέχρι το 2020 τα στοιχεία για τη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάρκοφ. Ήταν τεράστια αυτή, διάρκεια αρκετά αυτή η συνεδρίαση. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που έμειναν μέχρι τέλους. Ξέρετε κύριε Επίτροπε ότι ένας από τους συναδέλφους σας, τον οποίο δεν θα αναφέρω, ή μάλλον θα το πω, ο κύριος ε, Τίμερμανς δεν απαντά σε ερωτήσεις συναδέλφων που αποχωρούν από την αίθουσα. Εσείς απαντήσατε και ακόμα σε αυτούς που έφυγαν. Μπορεί να το ρωτούν περισσότερε ερωτήσει από ό,τι εμένα. Κανεί δεν ε, ερωτάται περισσότερο από εσά. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μα ενδιαφέρει το θέμα και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υπομονή τους και την προσαρμοστικότητά τους και το προσωπικό να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Επίτροπε που μας ενημερώσετε για το θέμα αυτό. Ε, πριν φύγετε συνάδελφοι να πω ότι θα συζητήσουμε τη δεύτερη δέσμη για τη διαλειτουργικότητα την οποία περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβριο αλλά θέλουμε να τελειώσουμε μέχρι το τέλος της θητείας. Ε, ήταν μακρά η συνεδρία, κουραστική για Δευτέρα απόγευμα, αλλά ήταν πολύ ε, ενδιαφέρουσα. Και είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι και να έχουμε και τις κατάλληλες απαντήσεις. Ε, να ευχαριστήσουμε λοιπόν και τον Επίτροπο και την ομάδα του που ήταν εδώ και τον επικεφαλής του Γιουλίσα και σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ. Ήταν ε, ένα κουραστικό απόγευμα Δευτέρας, αλλά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα λοιπόν και τους συναδέλφους που έμειναν μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ το εκτιμώ ιδιαίτερος και ορισμένες φορές κουράζεται κανείς ε, όταν έχει ταξιδέψει και την ίδια μέρα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την εισβάθος αυτή τη συζήτηση και να ευχαριστήσω και πάλι την ομάδα του Επιτρόπου και τον επικεφαλής του Γιουλίσσα. Ευχαριστώ.